Eh bien, bonjour et bienvenue. Καλημέρα σα, Καλώς ήρθατε. Θα ξεκινήσουμε την ημερήσια μάλλον την συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αντιρρήσει, σχόλια για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης υπάρχουν. Όχι. Άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έχετε λάβει τα πρακτικά της συνεδρίασης της 22 ε, Σεπτεμβρίου 2011. Αν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά, σας παρακαλώ να τα ανακοινώσετε στη γραμματεία μέχρι τη λήξη της συνεδρίασής μας. Η λήψη σχολείων παρατηρήσεων θα εγκριθούν τα πρακτικά. Με χαρά καλωσορίζω τους δύο βουλευτές ε, εθνικούς, τον κύριο Ζαν Πολ Μπακέ και τον κύριο Ζαν Λουί Κρίστα, οι οποίοι θα μας μιλήσουν ε, στη συνέχεια. Θα επανέλθω. Λοιπόν, άρθρο 192 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπει τις δραστηριότητες των συντονιστών των επιτροπών. Η αποφάση των συντονιστών πρόκειται, είναι κυρίως συστάσεις μέχρι ότου επικυρωθούν από την Επιτροπή. Μέχρι στιγμής ε, βασιζόμασταν στις πολιτικές ομάδες για να μας ε, ανακοινώσουν ε, πιθανές διαφωνίες των βουλευτών στις προτάσεις των συντονιστών η πρακτική διαβίβαση των αποτελεσμάτων ε, των συνδυάσεων των συντονιστών στα μέλη της Επιτροπής μέσω των πολιτικών ομάδων μέχρι σήμερα δεν μας ε, δημιούργησε κάποια δυσκολία. Ωστόσο, οι συντονιστέ προτείνουν από εδώ και πέρα τα αποτελέσματα των συνδυάσεων των συντονιστών να εγκρίνονται επισήμω με την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την έγκριση των πρακτικών των συνδυάσεων τη επιτροπή μα. Δηλαδή, Καταρχάς, έχουμε έγγραφο σχέδιο των αποτελεσμάτων της ε, συνεδρίασης των συντονιστών συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο των βουλευτών για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το σχέδιο των αποτελεσμάτων ε, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται αν δεν υπάρχει ε, κάποια ένσταση από τα μέλη της Επιτροπής μας που θα λάβει γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασης και τρίτον κατέτοιμα οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μπορεί να γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα αποτελέσματα της τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών που θα πραγματοποιηθεί στην συνδέση Επιτροπής στα διάφορα. Όταν τώρα εγκριθούν αυτά τα αποτελέσματα, επισυνάπτονται στα πρακτικά τη συνεδρίαση τη Επιτροπή, στη διάρκεια τη οποία εγκρίθηκαν. Συμφωνείτε να ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα αυτή τη διαδικασία. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε λοιπόν λάβει στο φάκελό σα τα αποτελέσματα τη συνεδρία των συντονιστών τη 22η Σεπτεμβρίου του 2011. Αν έχετε να διατυπώσετε παρατηρήσει σε σχέση με τα αποτελέσματα αυτά, σα παρακαλώ να τα αναφέρετε στη γραμματεία μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση. Αλλιώ εγκρίνονται τα πρακτικά. Τα αποτελέσματα μάλλον τη ε, της των συντονιστών. Δεν έχουμε ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη συνεδρία. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν έχω κάποια ανακοίνωση. Επομένως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσεις. Ο κύριος Ντομένικο Ρώσα, παρακαλώ, μήπως δεν είναι εδώ. Donc, il Άρα δεν υπάρχουν ανακοινώσει. Θέλει κάποιο το λόγο? Παρακαλώ. Πράγματι δεν είναι εδώ ο κύριος Νομένικο Ρώσα. Να σα πω ότι το πρόγραμμα εργασία 2012 της ΓΔ ε, και Αναπτυξής συνεργασία θα εγκριθεί την προσεχή εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, ωραία, το σημειώνουμε. Λοιπόν, τώρα περνάμε στα πιο επίσημα σημεία της σημερινής διάταξης. Ε, μπορούμε να φτάσουμε, μάλλον στα τα τυπικά το ολοκληρώσαμε και είμαστε στην ουσία. Είπα και πριν ότι με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τα δύο βουλευτέ τη Εθνική Γαλλική Συνέλευση, Ζαν Πολ και Ζαν Λουί Κρίστα, πρόεδρο και μέλο ε, τη ε, επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συγκεκριμένα. Υπάρχει μια ειδική αποστολή ενημέρωση, ο κύριο Μπακέ είναι πρόεδρό τη και στόχο είναι να ε, αξιολογηθεί η γαλλική πολιτική αναπτυξιακή βοήθεια και συγκεκριμένα την ισορροπία που πρέπει να εξεύρουμε σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθεια μεταξύ διμερών και πολυμερών προσεγγίσεων. Η συγκεκριμένη αποστολή ενημέρωση δημοσίευσε μια εντυπωσιακή έκθεση, παρουσιάστηκε στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τον Δεκέμβριο 2010 η αποστολή έθιξε διάφορα ζητήματα, τα οποία έχουμε και εμείς εδώ συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του μέλλοντος ε, της πολιτικής ευρωπαϊκής βοήθειας. Τα θέματα ήταν μεταξύ άλλων, ε, τα καλύτερα μέσα για την ενίσχυση του αντικτύπου της βοήθειας, το μεταβαλλόμενο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας και ρε, ρόλος των νέων χρηματοδοτών. Επίσης, η αποστολή στην έκθεσή της περιλαμβάνει υποδείξεις για το πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την καθοδήγηση των πολιτικών παροχής βοήθειας. Αυτό είναι πολύτιμο για τις συζητήσεις που έχουμε και εδώ στη δική μας Επιτροπή. Η έκθεση της αποστολής περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συνεργασία και ελπίζω ότι τις λεπτομέρειες αυτών των συστάσεων μπορούμε να τις συζητήσουμε μαζί σήμερα. Προτείνεται λοιπόν το ΦΕΔ να εγγραφεί στον προϋπολογισμό, κάτι που ζητάει άλλωστε εδώ και πολύ καιρό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντοτε άλλωστε υποστηρίζαμε την μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αλλά δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα δώσω αμέσως το λόγο στους Γάλλους συναδέλφους μου, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν αυτό που κατά την άποψή τους ε, συνιστά τη βασική, το βασικό συμπέρασμα της ε, έκθεσης της αποστολής τους. Λοιπόν, για 15 λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Μπακέ και ο κύριος Κρίστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Είχα την τιμή να προεδρεύσω στην ε, αποστολή τη διερευνητική αποστολή που διοργανώθηκε στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής σας για την αναπτυξιακή βοήθεια. Η Γαλλία είναι από τους πρώτους χορηγούς επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Βάσει του ΩΣΑ βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση πίσω από τη ΣΥΠΑ. Επίσης, 8 δις 900 εκατομμύρια καταγράφηκαν για το 2009 και κατά τι υψηλότερο ποσό για το 2010. Δεν δηλώνουμε ικανοποιημένοι παρόλα αυτά, ομόφωνα λυπούμεθα όλοι οι βουλευτές, διότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο το σύστημα, δεν επικρατεί διαφάνεια. Ε, δεν γίνεται κατανοητό το σύστημα και επίσης θεωρούμε ότι δεν επικρατεί ισορροπία. Δηλαδή η βοήθεια περνάει μέσα από συνεισφορές προς ε, πολύπλευρους οργανισμούς ή ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και λόγω αυτής της ανισορροπίας δεν έχουμε περιθώριο ελιγμών, ε, δεν έχουμε επαρκή επιρροή, ούτε προβάλλεται η εικόνα της χώρας μας ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό είναι το εφαλτήριο που οδήγησε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να οργανώσει αυτή την αποστολή. Για να συντάξουμε αυτή την έκθεση, φυσικά διάφορε εξέχουσε προσωπικότητε που ειδικεύονται στον τομέα συνεισέφεραν και κάναμε ε, στο Βιετνάμ, στην Τινησία, στη ΣΥΠΑ, στην Ελληνική Δημοκρατία του Κονγκό και στι Βρυξέλλε πέντε αποστολέ. Ε, καταδεικνύουμε έτσι το ενδιαφέρον μα ε, για να ακούσουμε τις χώρες που δέχονται αυτή τη βοήθεια, να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε για τα διάφορα εργαλεία συνεργασίας και να ακούσουμε επίσης την άποψη και άλλων εταίρων της Διεθνούς Αναπτυξιακής Βοήθειας, ε, κυρίως προέρχονται από πολυμερείς οργανισμούς ε, για να δούμε κατά πόσο ικανοποιούμε τις προσδοκίες και κατά πόσο κατά τη γνώμη τους είμαστε αποτελεσματικοί. Υπάρχουν διάφορες προβληματικές ανάλογα με τη χώρα. Κάτω από τη Σάχαρα, η Ασία, οι μεσογειακές χώρες αναδυόμενες σε μελλοντικά οικονομικά ε, σε μεσαίου μεγέθου ε, χώρε. Σε κάθε χώρα απαιτεί, διαφορετικού είδους ε, βοήθεια και άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Επίση, οι λοιπές αποστολές αποσκοπούσαν στην εξέταση τη πολυμερού δράση. Συναντηθήκαμε με του επικεφαλεί των διαφόρων διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, Πνίδο, UNICEF, Παγκόσμια Τράπεζα, Αμερικανική Τράπεζα παγκόσμια ανάπτυξη, διεθνέ Ομοσματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη ΣΥΠΑ συναντηθήκαμε επίση με τον αντίστοιχο Αμερικανικό Οργανισμό που εξαρτώνται από το δημόσιο τομείο εκπροσώπου του Κογκρέσου και ούτω καθεξής. Στι Βρυξέλλε. Ε, συναντηθήκαμε με την πρόεδρο τη Επιτροπή, ε, την κυρία Εύα Ζολή. Επίση, συστηματικά έχουμε επαφέ ε, σε διμερές, σε πολυμερέ επίπεδο για να μπορέσουμε κατά τη διαστολή να δημιουργήσουμε μια σφαιρική εικόνα για τη δική του άποψη περί τη κατάστασης και να καταγράψουμε τι ανησυχίε του. Εγκρίθηκε ομόφωνα στην, στο κοινοβούλιο μα η έκθεση και ενέχει τρία μέρη. Δεν πρόκειται να το παρουσιάσω διεξοδικά, διότι πιστεύω ότι έχετε λάβει ένα αντίτυπο. Στο πρώτο κομμάτι κομμάτι ε, κάνουμε έναν απολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας ε, και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει ιστορικώς πως να εξετάσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια προς όφελος ε, των αναγνωστών. Η αναπτυξιακή βοήθεια αυτή βασίζεται ταυτοχρόνως σε δύο πυλώνες σε όλες τις δυτικές χώρες. Πρώτον, διεθνής αλληλεγγύη βορράς-νότος, να επιβεβαιώσουμε δηλαδή ότι η έγκριση από τη Γενική Συνάλευση του ΟΗΕ του σχετικού ψηφίσματος που θεσπίζει την αναπτυξιακή βοήθεια συμβάλλει στην κατάργηση της ένδυας ε, εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω. Ε, χάρη στην αναπτυξιακή βοήθεια κρύονται οι προσπάθειες των δωρητών και ε, το 2010 επιβεβαιώθηκε η προσήλωση της διεθνούς κοινότητας προς την επίτευξη αυτών των στόχων και εντατικοποίηση των προσπαθειών. Δεύτερον, ο συντονισμός των εθνικών αναγκών και των διεθνών αναγκών. Ε, δεν έχει ακόμη σαφή, γίνει σαφής αποτίμηση και σήμερα βλέπουμε στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων τη αναπτυξιακή βοήθεια που κάνουν διάφορε χώρε ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού. Επίση, οι ραγδαίε αλλαγέ που χαρακτηρίζουν τη διεθνή σκηνή φυσικά επηρεάζουν ε, τις επιπτώσεις ε, της αναπτυξιακής βοήθειας και έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Επίσης, ο πολυμερή ή ο χαρακτήρα. χαρακτήρας τίθεται υπό αμφισβήτηση γιατί λόγω της παγκοσμιοποίησης υπάρχουν υπάρχουν ε, διάφορες, ε, παραδείγματος χάρη επιδημίες, ε, κλιματικές αλλαγές που συνεπάγονται ότι πρέπει να δώσουμε μια συλλογική απάντηση. Άρα χρειάζεται συνοχή ανάμεσα στα διάφορα όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας για να είμαστε αποτελεσματικοί στην αναπτυξιακή μας βοήθεια και να λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες των δικαιούχων. Έτσι σε διεθνές επίπεδο έχουμε αναλάβει διάφορες δεσμεύσεις είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο όπω παραδείγματο χάρη στο Μόντρε, στο Παρίσι το 2005 και δεν είναι τυχαίο που η G20 πλέον ε, ασχολείται με αυτό το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, όλα αυτά για να σας πω ότι η ανισορροπία ανάμεσα στο διμερή και πολυμερή χαρακτήρα της αναπτυξιακής βοήθειας που απασχόλησε αυτή την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μας είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή δεν επαρκεί να προσαρμόσουμε κατά τη προσπάθειά μας και να κλείνει η πλάστιγκα προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση για να λύσουμε το πρόβλημα. Μιλάω γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο, Πρόεδρε, αλλά Εντάξει, θα υπερβείτε το χρόνο σας. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν αλλαγές που επηρεάζουν και την διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια. Φυσικά η εξέταση του θέματος ε, από πλευράς μας όφιλε να λάβει υπόψη αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Ε, ο πολυμερής και διμερής χαρακτήρας αναπτυξιακής βοήθειας είναι μάλλον αλληλοσυμπληρωματικοί ε, και δεν βρίσκονται σε κανένα ανταγωνισμό. Για να είμαστε αποτελεσματικοί χρειαζόμαστε συλλογικές δράσεις στα πλαίσια της πελημερούς αναπτυξιακής βοήθειας ε, ε, και επανέρχομαι σε αυτά που σα έλεγα για τα ε, παγκόσμια δημόσια αγαθά για την καταπολέμηση επιδημιών κτλ. Κατόπιν, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι η δομή τη Γαλλική αναπτυξιακής Βοήθεια. Είμαστε από του βασικότερου χορηγού λόγω τη γεωγραφική κατανομής της αναπτυξιακής βοήθειας, του συνολικού όγκου τη βοήθεια, τη θεματική ενότητα που καλύπτει και το ρόλο που διαδραματίζει στον ευρύτερο διάλογο. Επίσης, η αναπτυξιακή μας πολιτική ε, παρουσιάζει διάφορε ιδιαιτερότητε σε σχέση με του άλλου εταίρου μα ε, και ανεξάρτητα από τα όσα διαμείβονται στη διεθνή σκηνή, αυτέ οι ιδιαιτερότητε που χαρακτηρίζουν τη γαλλική πολιτική ε, μα οδήγησαν και στην, στην ανάδειξη διαφόρων προτεραιοτήτων ω προ τα όργανα που χρησιμοποιούμε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. βλέπουμε ότι η αρχιτεκτονική του συστήματο ζητά καλύτερο συντονισμό επιτόπου, ότι δεν επαρκεί η πολιτική καθοδήγηση, δηλαδή τα δικά μα τα εργαλεία χαρακτηρίζουν αυτά καθεαυτά από μια ανισορροπία. Ε, ε, οι φιλοδοξίε μα απέχουν πόρο από την πραγματικότητα. Υπάρχουν αντιφάσεις οι οποίε βλάπτουν ε, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία αυτή της πολιτική. Η τα δάνεια ε, σε σχέση με τις ε, χορηγίες, παραδείγματος χάρη στις φτωχότερες, ε, έχουμε περάσει από τις φτωχότερες χώρες στις, αξιό, στις φερέγγιες χώρες. Αυτό ισχύει παραδείγματος χάρη στην Αφρική νοτίου της Σαχάρας, αυτά στον τομέα της υδροδότησης, των διαφόρων υποδομών και όλες αυτές οι επιλογές που έχουμε κάνει έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική μας ενισχύεται έτσι αυτή η ανισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στον πολυμερή και το διμερή χαρακτήρα της αναπτυξιακής βοήθειας. Επίσης, κατά τη διαστολή με την αναπτυξιακή πολιτική των εταίρων μας, ε, διακρίνουμε μια βασική διαφορά. Ε, ε, η ίδια η πολιτική μας που χαρακτηρίζεται από αυτήν την ανισορροπία, ο χαρακτήρα χαρακτήρας των βοηθειών, η ίδια η φύση δηλαδή της πολιτικής μας μας διακρίνει και αυτή πρέπει να διορθώσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής αναβαθμιστεί η αναπτυξιακή βοήθεια. Φυσικά έχουμε κάνει διάφορες εισηγήσεις για να επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε αυτό το πολυμερή και δημερή χαρακτήρα της αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει όμως να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία ότως ώστε να υποφεληθούμε τα μάλλα από αυτό το πολυμερή χαρακτήρα της αναπτυξιακής βοήθειας διότι ε, παρατηρούμε τις διάφορες ε, διεθνείς τάσεις ε, και πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μας. λόγω των τωρινών προκλήσεων θα πρέπει να συμμετάσχουμε πλήρως στην πολυμερή βοήθεια. Χρειάζονται καλύτερες απενδύσεις για να επιτύχουμε αυτό το ρόλο που καλούμε θα να διαδραματίσουμε και έτσι σε ευρωπαϊκό ή σε παγκόσμιο επίπεδο η Γαλλία θα έχει τη θέση που της αντιστοιχεί. Αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή, αν θέλουμε να προβάλλουμε περισσότερο την αδειξιακή μας σε βοήθεια. Θα πρέπει να βάλουμε σε τάξη τη διμερή αναπτυξιακή μα βοήθεια. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Ζαν Λουί Κρίστε, που με περισσότερε ακόμη λεπτομέρειε ε, θα σας παρουσιάσει την ανάλυση και τι προτάσει μας. Σα ευχαριστώ πολύ. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Κρίστε. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Θα συμπληρώσω τα λεγόμενα του συναδέλφου Ζαν Πολ Μπακέ και θα σας πω ακριβώς ποια είναι η συνέχεια σε αυτήν την αποστολή. Σας γνωρίζετε ότι η αναπτυξική βοήθεια πάντοτε εξάρτητα από το πλαίσιο, χθε ε, όπως και σήμερα αλλά και στο μέλλον στο διεθνές πλαίσιο, στο γεωπολιτικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζει την αναπτυξική βοήθεια και την εξέλιξη, επιλογέ τα εργαλεία, και το θέμα της αμνεξισορρόπησης των, θεσμικών, ε, των θεσμών ε, δεν ε, αποτελεί εξαίρεση. Η έκθεση λοιπόν για τις πολυμερείς και διμερείς σχέσεις που είναι και το εφαλτήριο του προβληματισμού μας επηρεάζεται άμεσα από την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και της θεματολογίας της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας. Λοιπόν, τα βασικά απορίσματα βασικά στηρίχθηκαν σε τρεις άξονες που ήταν διμερής προσέγγιση, ευρωπαϊκή προσέγγιση και πολυμερής προσέγγιση. Είναι λογικό ότι λαμβάνοντας υπόψη τις κριτικές ε, που έχουν ακουστεί για το σύστημα που ακολουθούμε, προσπαθήσαμε να δούμε το διοργανικό, το διαθεσμικό σύστημα στη Γαλλία και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε για να έχουμε καλύτερη πολιτική καθοδήγηση, μεγαλύτερη συνεκτικότητα και διευκρίνηση μεγαλύτερη των αρμοδιοτήτων. Στην Εθνοσυνέλευση λοιπόν ε, θα ε, πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις ορισμένα ζητήματα γιατί πράγματι έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρα όλα αυτά. Και όλοι οι παρατηρητές Μα ε, μας λένε και πρώτα απ' όλα στον ΟΣΑ ότι πρέπει να γίνει αυτό. Μεταξύ γάμα δέλτα ε, Δημοσίου Ταμείου και ΕΜΑΛ. Πολλές φορές σήμερα δεν ξέρουμε ε, ποιος είναι αυτός ο οποίος ορίζει και καθοδηγεί την πολιτική, την εξωτερική. Και βέβαια αυτό μπορεί να έχει επίπτωση και στις επιλογές και στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε. Και βέβαια είναι επιζήμιση ό,τι αφορά και την προβολή της πολιτικής μας. Το Γαλλικό Κοινοβούλιο από την πλευρά του θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει καλύτερα τις δημόσιες πολιτικές σε σχέση με, με τώρα. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι στη Γαλλία καμία συζήτηση δεν οργανώνεται υπό την αιγύδα της πολιτικής συνεργασίας δεν συμμετέχει στην έγκριση και την αναθεώρηση των τομεακών πολιτικών και των στρατηγικών. Βέβαια, μπορούμε να γνωρίσουμε ότι αρχίζει να αλλάζει λίγο η κατάσταση και είναι γεγονός ότι και η απαλλαγή ε, του Κοινοβουλίου είναι μια πολύ γαλλική παράδοση από το 1958 συγκεκριμένα, την Πέμπτη Δημοκρατία και είναι ένας από τους ε, λόγους για τους οποίους η περιθωριοποίηση του Κοινοβουλίου είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλει να... Ε, τι ισχύει με αυτή τη γαλλική παράδοση. Η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, πάνω απ' όλα, πώς να σας το πω, είναι ένα, μια ένα προνόμιο ε, για τον ε, πρόεδρο. Αυτή είναι η αποστολή ουσιαστικά που έχει. Ε, επομένως χρειάζεται μεγαλύτερη ειλικρίνηση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν κάποια αρνητικά στοιχεία τα οποία βλάπτουν την προβολή της πολιτικής που εφαρμόζουμε. Έχουμε επίσης μιλήσει, όπως σας είπα, ε, και για, το, για την εγγραφή του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό της αναπτυξιακής βοήθειας, ε, για να μιμηθούμε χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα και ακολουθεί αυτή την οδό δείχνοντας πόσο σημαντικές είναι οι διεθνείς δεσμεύσεις στον τομέα αυτό. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει επίση καλύτερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή πολιτική και συνεργασία, ώστε να γίνουν περισσότερο γνωστέ οι προσπάθειε και τα επιτεύγματα αυτή τη πολιτική και να συνεχίσει η κινητοποίηση στη χώρα μα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την εθελοντική ε, πολιτική στήριξη τη ε, ανάπτυξη και να φτάσουμε το επίπεδο άλλων χώρων. Πρέπει λοιπόν να προσελκύσουμε περισσότερο το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη. Ό,τι αφορά τώρα τι εταιρικέ σχέσει με τι δικαιούχου χώρε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ε, και αυτές μάλιστα οι χώρες ζητούν την προσέγγιση αυτή τις σχέσεις τους μεταξύ, ε, με τις δικές μας τις χώρες τη βλέπουν ακριβώς από αυτό το πρίσμα. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιωποιήσουμε και την χρηματοδότηση, να ε, διαρθρώσουμε καλύτερα τα διάφορα μέσα και εργαλεία και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας. Για να είμαστε λοιπόν πιο συνεπείς και συνεκτικοί, ζητήσαμε να υπάρξει σε βάθος προβληματισμός για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που θα πρέπει να οριστούν καλύτερα σε σχέση με τις ε, προτεραιότητές μας, γεωγραφικές και τομεακές. Μπορεί οι προσανατολισμοί ε, να ε, ορίστηκαν πρόσφατα και γενικές κατευθύνσεις και επιβεβαιώνονται και μετά τη δημοσίευση της έκθεσης πριν από ένα χρόνο περίπου. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά και την ε, Νοτιό Σαχάρα Αφρική, έχουμε ε, οι οποίες βλέπουμε ότι δεν ε, δεν έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε αυτή την πολιτική που θα την εξετάσουμε, την πολιτική των ενισχύσεων, την πολιτική των ε, δανείων. Θα πρέπει να, να θεωρώσουμε την προγραμματισμένη διμερή βοήθεια και να προσπαθήσουμε το 2015 να τη διπλασιάσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέσα αυτά, Σίγουρα είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλους ε, βασικούς ευρωπαίους χορηγούς και χρηματοδότες που μαζί με τις επενδύσεις τους, όχι τόσο στο ε, διμερές ε, σύστημα, έχουν κρατήσει μεν κάποια διμερή προγραμματική χρηματοδότηση και μπορούν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια σε χώρες ε, όπου εμείς δυστυχώς δεν έχουμε πολλούς πόρους και δεν είμαστε ούτε αποτελεσματική, ούτε προβαλόμεθα ιδιαίτερα. Ό,τι αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Συνεργασία και Πολιτική, και εσεί οι ίδιοι σίγουρα ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα γι' αυτά, τα ζητήματα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να μεγαλώσει η βαρύτητα ε, της Γαλλίας στο πλαίσιο αυτό. Η Γαλλία είναι μεταξύ των ιδρυτών του ΦΕΤ, του ΕΤΑ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη δηλαδή, και πραγματικά ε, πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να διαθρώσουμε καλύτερα του διάφορου τρόπου χρηματοδότηση, χωρί βέβαια σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσουμε τη δέσμευσή μα που κρατά εδώ και δεκαετίε. Το του λοιπόν. Είμαστε ο δεύτερος χορηγός του ΕΤΑ ήδη. Ε, δεν έχουμε την εντύπωση όμως ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία εκτιμά στη σωστή διάσταση τη συνεισφορά μας. Και σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, προσπαθήσουμε οι ε, υποσχέσεις και δεσμεύσεις της συνθήκης της Λισαβόνας να οδηγήσουν στην καλύτερη συμπληρωματικότητα και στην καλύτερη συνέργεια των πολιτικών συνεργασίας ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Έχουμε την πράσινη βίβλο της Κομισιόν και θέλουμε η Γαλλία να συμμετέχει πλήρως και να φροντίσει να γίνονται σεβαστές οι γεωγραφικές και τομεακές μας προτεραιότητες. Ταυτόχρονα ε, ζητούμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα ε, και στην δική μας την πολιτική, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ε, παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στηρίζοντας ε, τις ε, πολιτικές που ε, θα πρέπει βέβαια να συνάδουν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις πολιτικές των μεμονωμένων χωρών μέλων. ό,τι αφορά την εγγραφή του ΕΤΑ στο προπολογισμό, το είπε και ο Ζανπόλ φίλος και συνάδελφος, πρέπει να βρούμε τα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για μια διμερή πολιτική επιδοτήσεων στις στοχότερες χώρες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στα δάνεια της E Και θέλουμε να έχουμε μια σωστή, ε, μια σωστή προσπάθεια στην καταπολέμηση της φτώχειας. Και με τον τρόπο αυτό, με την εγγραφή του ΕΤΑ στον νομίζω ότι θα έχουμε ε, περισσότερα περιθώρια ελιγμών. Σε ό,τι αφορά τώρα το πολυμέρες σύστημα, καταλήξαμε σε ανάλογα συμπεράσματα Δηλαδή, είναι σημαντικό οι πολυμερείς οργανισμοί στους οποίους ε, συνεισφέρουμε να, γίνει σεβαστή, να γίνουν σεβαστές προτεραιότητές μας. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρχει ένα είδος αιρεσιμότητας ε, των ε, συνεισφορών, των συμμετοχών μας, ώστε να εξασφαλιστεί αυτός ο στόχος. Ο Σαν Πολμπακέ πολλές φορές ανέφερε τις ανισορροπίες που παρατηρούνται στο σύστημα δημιουργικής και θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές σε αυτό το επίπεδο. Πρώτα απ' όλα η εθελούσια συμμετοχή ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ δεν είναι επαρκής και θα πρέπει να ε, επανεκτιμηθεί αυτή η συμμετοχή. Συμφωνούν όλοι ε, και ευτυχώς αρχίζει να αλλάζει κάπως η κατάσταση. Επίσης, σίγουρα έχουμε εγκάρσια ταμεία Έχουμε το Παγκόσμιο Τόμιο για το Έτσι χάρη. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι παίζουμε έναν ρόλο πραγματικά επάξιο ε, των εισφορών που, που δίνουμε, ούτε σε ό,τι αφορά ε, και την πτυχή της ε, γαλοφωνίας, που δεν νομίζουμε ότι έχει τονιστεί επαρκώς. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα επί των οποίων είναι ευκταίο η Γαλλία να μπορέσει να τηρήσει καλύτερα τις δεσμεύσεις της και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τα διμερή εργαλεία και πώς μπορούμε να διαθρώσουμε καλύτερα ε, τα διμερεί. Εν κατακλείδη και εν συνόψη καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί πιο, ε, και να έχουμε μεγαλύτερη επιρροή. Παρ' όλα αυτά αυτό δεν συμβαίνει. Θα πρέπει να περάσουμε από συλλογικούς και πολυμερείς ε, μηχανισμούς λόγω αποτελεσματικότητας, ε, ανάγκης για μεγαλύτερη συνοχή, εταιρική ε, σχέση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα κάποια θέματα, να δούμε τη θεματολογία. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα, ούτε πρόκειται η Γαλλία να δεχθεί το να μειώνεται η προβολή της, η επιρροή της και ούτε βέβαια θα πρέπει να αλλοιώνεται, το, να αλλοιώνεται τα συμπεράσματα των εκθέσεων που δημοσιεύονται. Αντίθετα, βάσει και του επίπεδου βοήθειας ε, που παρέχουμε, έχουμε όλα τα όπλα στη διάθεσή μας ώστε ως Γαλλία να είμαστε σε ηγετική θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα ε, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να προωθήσουμε την και συνεργασία και τελικά να προσαρμόσουμε στα λόγια που λέμε τα έργα μας, δηλαδή τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και να τα κάνουμε πιο ε, ορατά και αποτελεσματικά. Και έτσι θα ξεκινήσει μια πραγματική δυναμική προ την εξέβρεση νέων εταιρικών σχέσεων. Κάτι το οποίο σήμερα είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Ευρωπαϊκέ στρατηγικέ, ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να γίνει για να ε, παγιώσουμε ακόμη καλύτερα το διμέρες και πολυμερές ε, σύστημα. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία ε, και σύζευξη αυτών των δύο πτυχών για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές Επιτροπής μας που επιθυμούν να, να σχολιάσουν. Ξεκινάς από την κυρία Κέλλερ. Um, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Με ακούτε. Ωραία και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι στην έκθεσή σας ε, τονίσατε την πολυμερή συνεργασία που πιστεύω πως έχει κρίση, σημασία καθώς είναι παγκόσμια το συμφέρον για την καταπολέμηση να πετύχουμε τους στόχους χιλιετίας κτλ. Και να πάμε ακόμη παραπέρα και αυτό είναι βεβαίω και στόχος και πολιτική διακήρυξη των ε, κρατών μελών ε, και της Ένωσης και του ΟΗΕ. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάτι το ωραίο και πολυμερές και έτσι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες αποτελεσματικότητας και συνεργασίας. Τότε χαίρομαι που πάτε σε αυτή την κατεύθυνση, παρά το ότι βεβαίως ε, δεν πειράζει να πάμε λίγο παραπέρα σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μια και μιλήσατε για τα συμφέροντα της Γαλλίας τα οποία θέλετε να διαφυλάξετε και να μην τα χάσετε ενώ συνεργάζεστε σε πολυμερές επίπεδο. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε ποια είναι αυτά τα μεγαλικά συμφέροντα. Και ένα πιο τεχνικό ερώτημα. Αυτή η αποστολή στην οποία πήγατε για πληροφόρηση τι ήταν ακριβώς. Ε, πρόκειται περί μια επιτροπής ad hoc που δημιουργήθηκε στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Να έκθεση αυτή πώς, πώς την κάνατε για όσου δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και μετά ένα ερώτημα για το πώ γίνονται, πώς αναπτύσσεται τι αναπτυξιακέ πολιτικέ στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Να το πούμε μετά αυτό ή όχι. Ή ευθύς αμέσως. No? Okay. Um, θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς αντιμετωπίζετε την αναπτυξιακή πολιτική στο Γαλλικό Κοινοβουλίο. Είπατε πως δεν έχετε πολλή επιρροή, αλλά πώς γίνονται τα πράγματα. Ε, εσείς επίσης που ασχολείστε με αυτό το θέμα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση με τους ε, συναδέλφους σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς συντονίζεστε, πώς φροντίζεται να υπάρχει μια συνοχή στην αναπτυξιακή πολιτική ε, γιατί βεβαίως αυτό μας απασχολεί πάντα εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να μάθουμε από εσάς κάτι πολύ ενδιαφέρον αν και βεβαίως δεν αφορά εσείς σας η οποία ούτως ή άλλως είναι πολύ ενδιαφέρουσα δεν ξέρω επίσης αν μας έχουν δώσει κανένα αντίγραφο ή τέλος πάντων κάτι μεταφρασμένο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. αυτό πολύ ενδιαφέρον. On va vérifier pour les copies, mais normalement... Θα το ελέγξουμε για τα αντίτυπα, αλλά κανονικά ένα λεπτάκι. D'accord. Alors on me dit qu'il existe uniquement en français, mais le με ενημερώνω ότι υπάρχει μόνο στα γαλλικά, αλλά υπάρχει η σύνοψη μέσα στο φάκελό σας. Ο κύριος ε, Γκέρινς τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τις δύο παρουσιάσεις. Η παρουσίαση του κυρίου Χρήστα με εντυπωσίασε περισσότερο, ομολόγο. Είπε, δεν ξέρουμε ποιο ακριβώ ε, προσδιορίζει στρατηγικέ επιλογέ, δηλαδή το ΙΠΕΞ ή ποιοι, ποιοι εταίροι, εν πάση περιπτώσει, αναπτυξιακή βοήθεια κάνουν στρατηγικέ επιλογέ. Μα είναι σοβαρό αυτό, έτσι ε, να μην ξέρουμε, να μην μπορούμε να εντοπίσουμε ποιο ε, κάνει τι στρατηγικέ επιλογέ. Δεν είναι προς τιμήν σας. Ε, διότι μπορεί να ε, ε, γίνουν όλα αυτά σε ένα ανώτερο επίπεδο, οι επιλογές δηλαδή. Εμείς στην αρχή της θετίας μας συμμετείχαμε στον προσδιορισμό αυτών των στρατηγικών επιλογών σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμό και συνοχή των πολιτικών, αλλά πώ να το καταφέρει κανεί αυτό, άμα δεν ξέρουμε ποιο έκανε τι στρατηγικέ επιλογέ. Ε, πρέπει να βάλετε τάξη σε αυτά. Αν ναι, εμείς οι βουλευτές ε, δεν ε, απευθύνουμε θερμή έκκληση για να γίνει κάτι, ποιος θα κινητοποιηθεί. Αναρωτιέμαι. Και αυτή είναι και η αχίλιος πτέρνα του ζητήματος για να απεμπλακεί η κατάσταση. Ε, κάνουμε γαργάρα διάφορες, ε, ε, διάφορα ευχολόγια για να λύσουμε το πρόβλημα της συνθήκης της Λισαβόνας, χωρίς όμως να λύσουμε τα ουσιαστικά προβλήματα που μας εμποδίζουν στο να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι θύνοντες. Euh, Κατόπιν, η πολυμερής και η διμερής διάσταση του ζητήματος. Ε, και πάλι εδώ θα πρέπει να δούμε ποιος κάνει στρατηγικές επιλογές και ε, θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε το θέμα σε λιγάκι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν έχουν επαρκές ειδικό βάρος ώστε μόλις έχουν πιστεί ε, για την καταλληλότητα των στρατηγικών επιλογών τους να καταφέρουν να τις ε, επιβάλλουν σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να είναι κανείς πεπισμένος για τις ε, δικές του επιλογές. Αν είναι, ε, θα πρέπει να τις προβάλλει και περισσότερο για να ακουστεί η φωνή τους στα διεθνή βήματα, μιλώντας για το αναπτυξιακό πρόγραμμα το ΙΕ. Εντάξει, ναι, συμφωνώ, αλλά Επίση και ε, στο πλαίσιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου τη Παγκόσμια Τράπεζα, γιατί και η Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί να κάνει λάθο. Ε, ε, στη ΦΑΟ Ε, στον Φάδο συζητούνται περίπου όλα τα θέματα, αλλά όταν ε, τους ε, ρωτάμε κάτι συγκεκριμένο, αν δηλαδή έχουν εξετάσει τις επιπτώσεις μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής επί της αναπτυξιακής βοήθειας, μας απαντούν ότι δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Υπάρχουν σαφέστατα κενά, αν θέλετε, και αδυναμίες στο πολυμερές διεθνές σύστημα. Τρίτη ερώτηση θα ήταν προς κοινό μας συμφέρον, πιστεύω, να εξετάσουμε ε, ε, αναλυτικότερα αυτό το θέμα και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο για το ζήτημα. Μήπως πρέπει να επαναπροσαρμόσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια στις ανάγκες των πλέον απόρων και με την Αραβική Άνοιξη θα πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά διάφορες δαπάνες μπορεί να είναι επιλέξιμες για την αναπτυξιακή βοήθεια ενώ κανονικά η βοήθεια διοχετεύεται αναδυόμενες χώρες ε, κατά κύριο λόγο. Για να σας τα πω σαφέστερα, για την Λιβύη νομίζω θα ήταν σκάνδαλο να επενδύσουμε ένα σέντ από την απτοεξιακή βοήθεια για να βοηθήσουμε τη Λιβύη. Έχει αρκετά χρήματα και δεν χρειάζεται ε, να χρησιμοποιούμε τα ήδη ε, ισχνά κονδύλια που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πείνα στον κόσμο για να βοηθήσουμε τη Λιβύη. Η Κίνα, η Ινδία που είναι αναδυόμενες ε, οικονομίες, η Κίνα έχει αναδυθεί, πάει, τελείωσε η, η βοήθεια που χορηγήθηκε βάσει των στόχων της αναπτυξιακής βοήθειας δεν πρέπει να σταματήσει. Άρα να επαναστοχοδετήσουμε τη βοήθειά μας. Τέταρτον, σωστά, τονίσατε τη σημαντική εισφορά της Γαλλίας στα πλαίσια της ε, διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας. Ε, σε, απο, ε, σε απόλυτους αριθμούς, εντάξει, αλλά υπάρχουν και σχετικοί αριθμοί, ξέρετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι πιστεύετε για την Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Αναπτυξιακή Βοήθεια. Θα ήταν πρόσφορο να μεταρρυθμιστεί το σύστημα κατά τη γνώμη σας, οι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί το 2005 συγκεκριμένα εξακολουθούν να είναι επίκαιρε. Ε, μια χώρα είτε ε, είναι μεγάλη είτε είναι μικρή, ε, αν ε, επιτύχει το 0,27% έχει ήδη επιτύχει το στόχο του ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια έτσι και ως προς την αναπτυξιακή πολιτική. Τώρα, σε σχέση με τις δωρεές ή τα δάνεια, την επιλογή ανάμεσα στα δύο, μήπως σταδιακά θα έπρεπε να απορρίψουμε την πολιτική δανειοδότηση σε όλες τις χώρες που έχουν προβλήματα διακυβέρνησης, διότι 20 χρόνια μετά την αντίστοιχη συμφωνία καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι πρόκειται για επισφαλή δάνεια, παραγράφουμε το χρέος και άρα το χρέος θα είναι και πάλι επιλέξιμο για τα ταμεία αναπτυξιακής βοήθειας, ε, τα κονδύλια δηλαδή που χορηγούνταν μέσα από αυτά τα ταμεία αναπτυξιακής ε, βοήθειας ήταν κονδύλια χαμένα, που πέφταν σε ένα απίθμενο πηγάδι. Μήπως ε, θα ήταν ε, πρόσφορότερο να ε, προτιμούμε τις δωρεές εξ αρχής από ότι να προσφεύγουμε διαρκώς στις, στους, στους ίδιους μαθηματικούς τύπους, στις ίδιες λύσεις μάλλον, που το καταδεικνύει η εμπειρία μας είναι μάλλον αμφίβολες. Ευχαριστούμε κυρία Γκέρενς. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο προς το παρόν, άρα... Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, όχι, δεν, δεν θέλετε. οι ε, κυρία Μπακέ και Κρίστας απαντήσουν ε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται για μια αποστολή ενημέρωσης. Αναφέρομαι στο ερώτημα της κυρίας Κέλλερ. Αποστολή ενημέρωσης λοιπόν του Γαλλικού Κοινοβουλίου που μπορεί να οργανώσει κοινοβουλευτικέ εξεταστικές επιτροπές όταν κάτι δεν φαίνεται ξεκάθαρο και αποστολές ενημέρωσης που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί κάτι. Και ενδεχομένως διατυπώνουμε και προτάσεις για βελτίωση του συστήματος. Άρα αυτή ήταν μια αποστολή ενημέρωσης. Για ποιο λόγο την οργανώσαμε αυτή την αποστολή ενημέρωση. Νομίζω ότι στα ερωτήματά σα, κυρία Κέλλερ, αλλά και στα ερωτήματα του κυρίου Βρίσκονται, βρίσκουμε ακριβώς τα στοιχεία της απάντησης, γιατί οργανώσαμε αυτή την αποστολή. Πώς λειτουργεί τώρα, ε, ποιος είναι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων, ε, ποιος αποφασίζει τι. Αυτά ήταν τα ερωτήματα τα οποία έθεσε και η Γαλλική Βουλή. Και δεν είναι λήψη απαντήσεων. Μάλλον και επειδή δεν είχαμε απαντήσεις, γι' αυτό και συγκροτήσαμε αυτή την αποστολή. Τώρα, ποια είναι τα συμφέροντα της Γαλλίας, μας ρωτήσετε κυρία Κέλλερ τι ακριβώς υπονοείται. Εμείς δεν υπονοούμε, ε, λέμε ξεκάθαρα. Η Γαλλία σήμερα, όταν είναι εντελώ αδιαφανές στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, είτε είναι διμερής, είτε είναι πολυμερής, και κάποιες φορές ε, ανεξέλεγκτη μη ελεγχόμενη, δεν αποκομίζει το όφελος τις βοήθειες που παρέχει. Όταν λέμε όφελος μπορεί να είναι η γαλλική σημαία, η ευρωπαϊκή σημαία. Είναι ένα είδος πολιτικής επιρροής η αναπτυξιακή βοήθεια. Κάποιες χώρες, είχα συναντήσει εδώ την κυρία Εύα Ζολή, η οποία μας είχε πει στο τέλος της συνεδρίασης τότε, δεν έχουμε το δικό σας πρόβλημα, γιατί εμείς οι Νορβηγοί δεν είμαστε ποτέ απεικιοκράτες. Είναι προφανές ότι απεικιοκρατικές χώρες πάντοτε και οπουδήποτε επιζητούσαν να έχουν προνομιακές σχέσεις με τις πρώην απικίες. Είτε λόγω μετάνοιας, είτε γιατί χρειαζόταν πλέον να δοθεί τότε που δεν είχε δοθεί και το χρωστούσαν στη χώρα αυτή. Υπάρχει όμως ε, μία μη αμεληταία πολιτική σχέση και αυτό αποδεικνύεται και το έλεγα και πριν με την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Προσωρινά τότε περάσαμε από έναν ε, διπολικό σε έναν πολυπολικό κόσμο. Είδατε τα στοιχεία για το κόστος αναπτυξής βοήθειας να καταρρεύουν σε όλες τις χώρες. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου βλέπουμε να αυξάνεται και εκ νέου η αναπτυξιακή βοήθεια. Βέβαια, πίσω από την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας, θα μου πείτε, υπάρχουν γεωστρατηγικές, γεωπολιτικές επιλογές. Και στις επιλογές αυτές υπάρχουν και κάποια στοιχεία ασφάλειας, καθόλου αμεληταία. Η εταιρική σχέση της Γαλλίας δεν έχουμε σκέψεις ε, από πίσω, είναι ξεκάθαρα όλα. Υπάρχει όμως και αυτή η λέξη εταιρική σχέση, κάτι καινούριο. Και επιμένουμε σε αυτό στην έκθεσή μας. Η αναπτυξιακή βοήθεια, και το εξηγούμε στην αρχή της έκθεσης, ε, τη γέννηση δηλαδή της έννοιας της αναπτυξιακής βοήθειας στη Γαλλία, που την κληροδοτήσαμε από μια χριστιανική παράδοση αλληλεγγύης ουσιαστικά και από τη νεοαπικιοκρατική ίσως προσέγγιση η Γαλλία της Αφρικής. Θα έχετε ακούσει να γίνεται λόγος για αυτή την έκθεση, Ανάγκη μετά να αλλάξουμε τελώς τα πράγματα. Και από τη στιγμή που θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να έχουμε δύο εταίρου. Άρα η αντεξική βοήθεια μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο μια εταιρική σχέσης. Δεν αποφασίζει αυτός που χορηγεί μόνο. Είναι η εταιρική σχέση αυτή που εγκαθιδρύεται μεταξύ του δωρητή και του δικαιούχου και του αποδέκτη. Ένα τελευταίο τώρα σχόλιο για την πολιτική διάσταση. Πράγματι το λέει και στην έκθεσή μας, όταν λίγα λέει ότι θα πρέπει ε, να επικεντρώσουμε τη βοήθειά μας γεωγραφικά και κυρίως στην νοτέως της Σαχάρας Αφρική, αυτό το κάνουμε γιατί μιλάμε για μια πολιτική εγκύτητας. Είναι προφανές αυτό. Δεν είναι διαφανής η βοήθεια σήμερα, είναι διάχυτη η βοήθεια αυτή και πολλές φορές ε, δεν τελείπω κανέναν έλεγχο. Και σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του κ. Γκέρενς, να πω ότι πράγματι η πρόταση που κάνετε εσείς ε, είναι και στην έκθεσή μας. Δηλαδή να προτιμηθούν οι δωρεές σε σχέση με τα δάνεια. Δηλαδή οι φτωχότερες χώρες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δάνεια, που δεν μπορούν και να τα αποζημιώσουν, κινδυνεύουν να γίνουν φτωχότερε ακόμη χώρες και να μείνουν τελείως εκτός πορείας ε, ανάπτυξης. Ακριβώς γι' αυτό κάνουμε και αυτή την πρόταση που κάνατε κι εσείς. Ευχαριστώ. Μάλιστα, για να συμπληρώσω αυτά που μας είπε ο κύριος Μπακέ, θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, ε, σε σχέση με την ε, δυσκολία που έχουμε για να γίνει κατανοητό το σύστημα ακόμη και στα δικά μας ε, θεσμικά όργανα, κάναμε διάφορες εισηγήσεις, μεταξύ των οποίων και μια πρόταση για να βελτιώσουμε γενικότερα το μηχανισμό και να γίνει καλύτερα κατανοητό. Προτείνουμε μεταρρύθμιση τη αρχιτεκτονική του σύστημα, ώστε να καταστεί δυνατή μια αναβαθμισμένη πολιτική καθοδήγηση. Ε, για να επιτύχουμε αυτό το στόχο θα πρέπει να εμπλακεί σε μεγαλύτερο βαθμό ε, τα, το κοινοβούλιο κάθε χώρα. Οπότε προτείνουμε να εγκριθεί ένας νόμος ε, πλαίσιο για την αναπτυξιακή πολιτική της ε, Γαλλίας, να διοργανώσουμε μια, ένα ετήσιο διάλογο, μια ετήσια εξέταση του θέματος επί τη βάση της έκθεσης που θα μας υποβάλει η κυβέρνηση κάθε χρόνο. Εμπλέκεται λοιπόν το κοινοβούλιο καθώς και για την υιοθέτηση των τομεακών πολιτικών στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η πρότασή μας ε, και θα θέλαμε να υλοποιηθεί ε, ούτω ώστε να εμπλακεί σε μεγαλύτερο βαθμό λοιπόν το κοινοβούλιο. Ε, η ερώτηση τώρα που θέσατε για την συνένεση, την ευρωπαϊκή συνένεση, προφανώς ε, ε, στις προτάσεις μας αυτό επιδιώκουμε και εμείς πάντοτε, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, μεγαλύτερη διαφάνεια για την αναπτυξιακή πολιτική, να διατηρήσει το 0,7% γιατί έχουμε αναλάβει διεθνείς δεσμεύσεις, αλλά όχι μόνο, στα πλαίσια του, του ΓΚΑΤΕ έχουμε και άλλες δεσμεύσεις ε, πάλι στα πλαίσια της αναπτυξιακής ε, βοήθειας, ε, οπότε... Δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για τους αριθμούς και ούτως ή άλλως χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτά. Α, ναι, και κύριε Γκέρενς, όταν αναφερθήκατε σε διάφορες σχέσεις που υπάρχουν, κοιτάξτε, καλό θα ήταν εδώ να σκιαγραφίσουμε μια πιο δραστήρια, αν θέλετε, εταιρική σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να βάλουμε από κοινού όλα τα μέσα που διαθέτουμε, να υλοποιήσουμε κοινέ στρατηγικέ, ούτω ώστε να είναι πραγματικά αποτελεσματική η βοήθεια. Ταυτόχρονα, μια σοβαρότατη έλλειψη είναι η εξή. Ε, δεν υπάρχει επικοινωνιακή πολιτική ε, προ του πολίτε μα, ε, όχι σε επαρκή βαθμό για να του καταδείξουμε με ότι γίνεται ευλογή ε, χρήση της ε, βοήθειας. Θα αναφέρατε κι εσείς ότι έχει κέρια σημασία η καταπολέμηση της ε, ενδίας, αλλά νόημα έχει μόνο αν μεριμνήσουμε ώστε όλοι αυτοί που εκπροσωπούμε να προσχωρήσουν σε αυτήν τη στρατηγική. Χρειάζεται λοιπόν πραγματική επικοινωνιακή πολιτική και ε, θέση από κοινού όλων των μέσων που διαθέτουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και ελπίζουμε με αυτές τις προτάσεις που ακούσατε να ξεκινήσετε κι εσείς μια αντίστοιχη διαδικασία και κυρίως να επιτύχουμε μεγαλύτερη συνεργασία για τα αναπτυξιακά ζητήματα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Κυρία Ατού. Euh, Σας ευχαριστώ. Είμαι από τη Γαλλία, είμαι μέλο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Επιτροπή Ανάπτυξη. Είπατε, κύριε Κρίστο, ότι και παράπονο σε αυτό που είπατε, θα πρέπει να διαπρατευτούμε με τι διάφορε χώρε και ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί κάποιε φορέ δεν κάνουν αυτά που πρέπει. Έχω την εξή ερώτηση προ εσά. Αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που έχουν γίνει, με τον άνεμο εκδημοκρατισμού που πνέει, μήπω θα ήταν ώρα να ξαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει όχι μόνο με τι χώρε ε, και δει με, ε, με καθεστώτα πολιταρχικά, ε, αλλά με το λαό, όχι με τι κυβερνήσει που δεν είναι και νομιμοποιημένε, με το λαό να γίνει διαπραγμάτευση. Να έχουμε χρόνο να διαπραγματευτούμε με το λαό πλέον και όχι τη χώρα που δεν είναι δημοκρατική. Ας δούμε τι έγινε με τη Λιβύα και την Τινησία. Με τη Λιβύα και την Τινησία διαπραγματευτήκαμε τον Καντάφη, διαπραγματευθήκαμε με τον Μπεναλή. Αλλά δεν ακούσαμε και το λαό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν κατά την άποψή σας για να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι η προτεραιότητα σήμερα είναι η νοτίος της Σαχάρας Αφρική. Αλλά Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλέ κυβερνήσει, πολλοί πρόεδροι σε χώρε τη Ποσχάρη Αφρική ε, δεν εκπροσωπούν το λαό του, το λαό τη χώρα του. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε να διαπραγματεύσουμε πολιταρχικού ε, ηγέτε. Αν λοιπόν θέλουμε ο λαός να βγει από τη φτώχεια, αν θέλουμε να έχουμε διαπραγματεύσεις με κυβερνήσει μη νομιμοποιημένε και απολυταρχικέ, δεν γίνεται. Πριν από κάποια χρόνια Είχα συναντήσει έναν τώρα υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών ε, της Γαλλίας και μου είχε πει «Α, ναι, εσείς είστε αυτοί που ασχολείστε με τα ανθρώπινα δικαιώματα». Και το είχε πει κάπως υποτιμητικά, επιτιμητικά. Μα ξέρετε, δεν μπορούμε να ακούμε τις κυβερνήσεις μόνο, πρέπει να ακούμε και τους λαούς των χωρών αυτών. Πώς θα το πετύχουμε. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να σας πω όμικρον, κυρίω από αφρικανικέ χώρε που εργάζονται για τα θέματα αυτά και που θέλουν να φύγουν οι χώρε, ε, οι λαοί των χωρών αυτών από τη φτώχεια. Άμα σα πούνε ότι δεν σα θέλει, δεν θέλουμε αυτή την αναπτυξιακή ε, πολιτική, θέλουμε μια ισότιμη σχέση. Θέλουμε να καταβάλλετε δίκαιες τιμές για τους φυσικούς μας πόρους και δεν θέλουμε να νιώθουμε ότι εσείς έχετε ένα αίσθημα ανωτερότητας απέναντί μας, ότι μας βλέπετε αφιψηλού. Μπορεί μήπως πλέον αυτή η σχέση η αναπτυξιακή να αντικατασταθεί από μια ισότιμη σχέση με χαρακτηριστικά ισότητας και αδελφοσύνης. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κρίστη να απαντήσει. Θα έρθω σε αυτό που είπατε. Ε, αναφέροντας τελευταία μας λέξη, εταιρική σχέση. Αυτό ήταν και το αντικείμενο τη διάσκεψη κορυφή τη Λισαβόνα. Ευρώπη-Αφρική, εγκαθίδρυση μια νέα εταιρική σχέση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα των πολιτικών που ακολουθούμε σήμερα. Να έχουμε μια ισότιμη ε, σχέση. Ίσως προ ίσον. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια δυσκολία. Έχουμε κάποια καθεστώτα ε, που δεν ξέρουμε πώς να τα χειριστούμε. Και έχουμε εδώ εμείς ε, καθιερώσει μια διπλωματική, μια κοινοβουλευτική διπλωματία. Δηλαδή να συναντηθούμε με κάποιους βουλευτές, ε, να ε, δημιουργήσουμε επικοδομητικές σχέσεις που θα μας επιτρέψουν να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, να δούμε ποιος είναι ο δημοκρατικός μηχανισμός, το δημοκρατικό σύστημα που ισχύει σε κάποιες χώρες. Πάντοτε θέλουμε και το λέμε να ξεκινήσουμε ε, σχέσεις με πολιτικούς, γιατί πολιτικοί είμαστε. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική διπλωματία νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθεί. Και υπάρχει και ένα άλλο σύστημα, ένας άλλος μηχανισμός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αλλαγή και στην βελτίωση των ανταλλαγών. Είναι η αποκεντρωμένη συνεργασία. Η αποκεντρωμένη συνεργασία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπει από τη μια πόλη στην άλλη, από μια ένωση σε μια άλλη ένωση να δημιουργηθούν αυτές οι σχέσεις ε, Συμμετοχή παραδείγματο χάρη στο κράτο δικαίου. Ξέρουμε ότι το κράτο δικαίου είναι στόχο, είναι στόχος ε, των στόχων της ε, χιλιετίας, για παράδειγμα, των αναπτύξεων στόχων τη χιλιετίας και πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, αλλά θα ήταν λίγο αφελές να πιστεύει κανεί ότι μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να δημιουργήσουμε τέτοιε σχέσει με τον, ε, αν το δει α με τη ε, την Επανάσταση, ο λαός τη ε, αντέδρασε. Και αυτή η όθηση του λαού τη Τινησία ήταν αυτή η οποία οδήγησε ε, στην δημοκρατική αυτή προσέγγιση και πορεία στη χώρα. Μόνο έτσι μπορεί λοιπόν να ε, επιτευχθεί πρόοδος. Ε, σίγουρα υπάρχει ανάγκη να γίνει η αλλαγή με κάποια καθεστώτα που εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά δεν αλλάζουν τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Παραλαμβάνω, κοινοβουλευτική διπλωματία μπορεί να βοηθήσει οι σχέσεις αυτές που οικοδομούνται μέσω των πόλεων, η αποκεντρωμένη συνεργασία. Δεν είναι εύκολο, αλλά ίσως είναι πιο εύκολο να εκφράσει κανείς έτσι την απληπισία, την απόγνωση, την κριτική του, παρά να δημιουργήσει έναν αυθεντικό μηχανισμό και σύστημα. Δεν υπάρχουν κανόνες. Πώς να το πω, ε, δεν υπάρχει ε, κάποια δυνατότητα από τη μια στιγμή στην άλλη να υπάρξει τροποποίηση αυτών των απολυταρχικών καθεστώτων αυτόματα, δεν υπάρχουν τόσο εύκολα εργαλεία όπως ε, τουλάχιστον εσείς ε, δείχνετε να πιστεύετε για να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Αλλά επαναλαμβάνω, μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, μέσω μιας ε, πολιτικής αποκεντρωμένης συνεργασίας, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτά τα καθεστώτα. Euh, Επιτρέψτε μου να προσθέσω κι εγώ κάποιες σκέψεις. Έχετε δίκιο, κάποιες χώρες αρνούνται τη βοήθεια. Έχετε διαβάσει σίγουρα ένα βιβλίο που ονομάζεται «Η μοιραία βοήθεια». Ε, τι εννοούμε όμω όταν μιλάμε για εταιρική σχέση. Ε, σημαίνει ότι ε, επί ίσης συζητούν οι δύο εταίροι. Δηλαδή για μακρά χρονική περίοδο τι κάναμε. Είχαμε αποφασίσει εμείς ότι θα τρέξει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν σημαίνει αυτόματα ότι παρουσίαζε κάποιο όφελος για την δικαιούχο χώρα. Ε, και το κάναμε για να, μας, ε, ε, για έχουμε την επιστροφή, την απόσβεση για τις επενδύσεις μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Εμείς επιδιώκουμε μια πραγματική ουσιαστική εταιρική σχέση στο Βιετνάμ παραδείγματο χάρη με όλη τη δουλειά που κάνει η αντιπροσωπεία μας εκεί, στο Ανόη λοιπόν, Τώρα δεν, μπορώ δεν μπορείτε να με αναγκάσετε να σα πω ότι πρόκειται για δημοκρατικό καθεστώ, αλλά τέλο πάντων δεν έχει σχέση αυτό. Είχαμε ενώπιόν μα εταίρους που κάποια πράγματα τα δέχτηκαν, κάποια τα αρνήθηκαν. Δηλαδή αξιολογούσαν, βλέπανε ποια δράση παρουσιάζει κάποιο συμφέρον για εκείνους και το δέχονταν και επίση. Βλέπαμε, βλέπανε ε, ε, ότι υπήρχαν κάποια προγράμματα που δεν προσαρμόζονταν στι ανάγκε, του παρότι εγγράφονταν στα πλαίσια τη δική μα εθνική πολιτική. Ήταν υπεύθυνοι λοιπόν και σας, ε, ε, υπό αυτές τις περιστάσεις ε, ξέρετε προς τα που οδεύετε και αυτό είναι πολύ καλύτερο δηλαδή μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον για άλλους αυτή, ε, αυτή ήταν η πρώτη σκέψη δεύτερη σκέψη είπατε ότι πρέπει κάποιος να πληρώσει την εύλογη τιμή τη σωστή τιμή ε, κοιτάξτε, τώρα πρόκειται για μια άλλη πρακτική της αναπτυξιακής βοήθειας, αναπτυξιακής εισαγωγικά, γιατί δεν φέρνει ανάπτυξη, πρόκειται για λαιλασία. Ε, έρχονται κάποιοι για να σας φτιάξουν ένα στάδιο ε, ε, ε, ποδοσφαιρικό, επειδή τους έχετε παραχωρήσει για 25 χρόνια την εκμετάλλευση κάποιου ορυχείου. Συγγνώμη, αλλά δεν πρόκειται για ανάπτυξη. Και όπως ε, είπαμε, είπανε και άλλοι, για μια σωστή εταιρική σχέση χρειάζονται ε, δύο εταίροι. Μπορεί να μην είναι, ε, δεν πρόκειται για τα πολιτικά καθεστώτα που επιθυμούμε εμείς, αλλά να μην είναι τουλάχιστον εντελώς διεστραμμένα, να μην στραγγαλίζουν τον ντόπιο πληθυσμό. Πρέπει να έχουμε επίγνωση όλων αυτών. Τρίτον, σε σχέση με αυτά που έλεγε ο συνάδελφος, ε, για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Βεβαίω, πολύ ε, καλό. Ε, θα πρέπει να εμπλακούν οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές γιατί ξέρετε ότι δεν μπορεί να μετεξελιχθεί ένα σύστημα δεν γίνεται κατανοητό. Δεν μπορεί πίσω από την πλάτη της χώρας να τα κάνουμε αυτά. Πρέπει να δεχτούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους... Γι' αυτά σα μιλούσα προηγουμένως... Δηλαδή, στην κρίση που βιώνουμε τώρα υπάρχουν ε, κάποιοι που υποφέρουν, που πλήττονται και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν είμαστε σε περίοδο μεγάλη οικονομική ανάπτυξη ε, και κυρίως σε περίοδο κρίση ε, χρειάζεται κατανοητή γλώσσα για να καταλαβαίνουν όλοι περί πρόκειται. Και λοιπόν η αποκεντρωμένη συνεργασία, είναι κέριο εργαλείο για να καταλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, και αντίθετα με αυτό που μας είπε ο συνάδελφος, ε, θα, δεν θα επιθυμούσα πλήρη αποκέντρωση, θέλω ένα μικρό βαθμό συγκέντρωσης. Ε, δεν γίνεται να πηγαίνουν στο, στην Πούρκινα Φασό, στο Μαλί και στο Νίγηρα ε, όλα τα λέει και να ξεχνάμε όλες οι υπόλοιπες χώρες. Εντάξει, αυτές είναι εύκολες οι χώρες. Ξέρουμε, ξέρουμε ότι εκεί πέρα επικρατεί μιζέρια. Γνωρίζουμε τις ανάγκες αυτών των ε, χωρών και να είναι αποκεντρωμένη η βοήθεια. Συμφωνούμε και εμείς, αλλά νομίζω θα ήταν χρήσιμο ε, να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο σε ένα μικρό βαθμό να διαχειρίζεται ε, κεντρικά η αναπτυξιακή βοήθεια. Ένα μικρό ποσοστό και το μεγαλύτερο ποσοστό να αποκεντρωθεί. Ε, αυτό είναι μεταξύ των προτάσεών μας. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Δεν ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι τους κυρίους Κρίς και Μπακέ που ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω πραγματικά ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια στενότερη συνεργασία με το Γαλλικό Κοινοβούλιο. Όπως ξέρετε, ήδη από αύριο το απόγευμα έχουμε διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με το Γαλλικό Κοινοβούλιο για την αιρεσιμότητα της ε, βοήθειας ε, ως προς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε και αν θέλετε να παραμείνετε φυσικά είσαστε ευπρόσδεκτοι. Διακόπτουμε δύο λεπτά. Πολύ ωραία. Θα περάσουμε τώρα στην παρουσίαση από πλευρά τη κυρία Λέβιν. Δεν ξέρω, πότε δεν ξέρω, πώ παραφθείρω το όνομά σα. Όχι, ωραία το είπα. Λέβιν, για το σχέδιο γνωμοδότηση για την Επιτροπή Αλία σχετικά με ε, τη Συμφωνία Λευτικής Σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου. Το Κοινοβούλιο καλύτερα να εγκρίνει να απορρίψει την σύναψη αυτή της ε, συμφωνίας. Έχετε το λόγο κυρία Λέβεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήρθα τρέχοντας από την Επιτροπή Αλληλείας όπου συζητούσαμε ακριβώς το ίδιο θέμα με τον εισηγητή της ε, Άλντε. Να σας δώσω εδώ πέρα το ιστορικό στην Επιτροπή σας. Η πρώτη συμφωνία αλληλευτική με το Μαρόκο υπεγράφει το 1995. Το καιρό εκείνο ήταν η πιο σημαντική αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτης χώρας. Όμως τα μέρη δεν έφτασαν σε συμφωνία ανανέωση του πρωτοκόλλου το 1999, οπότε δεν υπήρχε μια συμφωνία μέχρι να τεθεί εν ισχύ η φυστάμενη αυτή συμφωνία του Φεβρουάριου του 2007. Και το πρωτόκολλο αυτό βεβαίως είχε τετραετή ισχύ, εξέπνευσε τον Φεβρουάριο φέτος, οπότε αυτό το οποίο συζητάμε τώρα είναι μια προσωρινή παράταση της συμφωνίας αυτής και βεβαίως αυτή η προσωρινή παράταση ε, αντικείμενο γρήγορη διαπραγμάτευση από την Κομισιόν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο φέτος και να σας πω το γιατί συζητάμε τώρα μόνο προσωρινή παράταση του πρωτοκόλλου τον Μάιο του 2009 η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Ανάπτυξης ε, ζήτησε μια γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για την νομιμότητα της συμφωνίας αυτής καθώς καλύπτει και τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Η Δυτική Σαχάρα είναι μια επικράτεια η οποία δεν έχει αυτοδιοίκηση την οποία θεωρεί όμως τμήμα του το βασίλειο του Μαρόκου, κάτι το οποίο ποτέ δεν έχει αναγνωριστεί από τον λαό της Δυτικής Σαχάρας και τους αντιπροσώπους του και από τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεν έχει καν ορίσει το Μαρόκο ως την ε, διαχειρίστρια δύναμη της ε, Δυτικής Σαχάρας, παρά μόνο ως την χώρα η οποία de facto διαχειρίζεται τη Δυτική Σαχάρα. Σύμφωνα με κάποια ψήματα του ΟΗΕ και της απόφαση ε, του Συμβουλίου Ασφαλείου του 1992 θα έπρεπε να έχει υπάρξει ένα δημοψήφισμα για να μπορέσει ο λαός να εκφράσει το δικαίωμά του στην αυτοδιάθεση του ή όχι. Αλλά βεβαίως δεν έχει διεξαχθεί κανένα δημοψήφισμα καθώς δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία. Περιτώ να σας πω πως ο λαός της ε, Σαχάρας ή Σαχαράουι βεβαίως ε, ε, υφίσταται έναν επικισμό από Μαροκινούς, τους οποίους πλέον προσελκύει η η εκεί πέρα με χαμηλό το καδάνια και πλέον οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται ντόπιοι. Οπότε το ερώτημά μας ήταν εάν η συμφωνία αυτή στην οποία με την οποία θα έχουν πρόσβαση οι αλληλείς Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ύδατα της ε, Διεθνούς Σαχάρας ε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Και ε, το 2001 απάντησε η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου και το εξηγήσαμε και η απάντηση ήταν όχι. Βασίστηκε η νομική υπηρεσία στη γνωμοδότηση του Χάντ Κορέλο, ο οποίος ήταν νομικός συμβουλός του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία η αδίποτε δραστηριότητα έρευνα ή εκμετάλλευση της Δυτική Σαχάρα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον είναι προ όφελο και σύμφωνα με τις επιθυμίες του λαού της δυτική Σαχάρα. Και η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέτασε τη συμφωνία αυτή, όλα τα νούμερα, τα στοιχεία, τα έγγραφα που έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν βρήκαν ε, κάποιο στοιχείο σύμφωνα με το οποίο η συμφωνία αυτή είναι προς όφελος ε, ή σύμφωνα με τις επιθυμίες του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Και άρα η νομική υπηρεσία αυτού του Κοινοβουλίου συνέστησε να ανασταλεί ή να επαναδιαπραγματευτεί αυτή η συμφωνία αποκλείοντας τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας αυτή τη γνωμοδότηση παρουσιάσαμε και στην Επιτροπή Αλίας. Η Κομισιόν δέχτηκε πάρα πολλές ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές και εν μέρη λόγω αυτής της πολιτικής πίεσης η Κομισιόν άρχισε να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στο Μαρόκο. Το εάν αυτή η συμφωνία λοιπόν ωφελεί τον πληθυσμό τον τοπικών Οι του Μαρόκου δεν απάντησαν, υπήρχε μία προθεσμία που ήταν Αύγουστος του 2010 και ανέμενε μια απάντηση η Κομισιόν για να μπορέσει να αξιολογήσει το εάν αυτή η συμφωνία ήταν σύμφωνη προς το Διεθνές δίκαιο ή όχι. Για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία όταν έληξε το πρωτόκολλο τον Φεβρουάριο. Αλλά το Μαρόκο δεν υπέβαλε καμία απάντηση μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου πέρσι. Δύο μήνες πριν τη λήξη της συμφωνίας. Και τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν ήταν πολύ επιφανειακά. Τα έχω δει. Είναι μια παρουσίαση PowerPoint και μπορείτε να τα βρείτε στο site της γραμματείας οπότε φαντάζομαι μπορεί να το δουν όλοι οι ευρωβουλευτές και περισσότερο περιγράφει την αλληλευτική πολιτική του Μαρόκου και δεν είναι βεβαίως αξιολόγηση της συμφωνίας αυτής δεν αναφέρει καν τη δική Σαχάρα μόνο πολύ επιφανειακά αναφέρει κάποιες επενδύσεις που έγιναν στο Μαρόκο. Τίποτα άλλο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση αυτά ζήτησε μία παράταση του πρωτοκόλλου για ένα έτος προσωρινή παράταση για να μπορέσει η Κομισιόν να αξιολογήσει τα γεγονότα αυτά και να δει το τι θα γίνει με την αληφτική αυτή συμφωνία. Η Επιτροπή Αλληλείας απογοητεύτηκε πάρα πολύ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η συγγήτρια η οποία έχει οριστεί έχει τη μόνη έκθεση αξιολόγηση της προηγούμενης ε, συμφωνίας ε, την οποία έκανε ένας ανεξάρτητος σύμβουλος που κανονικά κάνει αυτά τα πράγματα και το έλαβαν μόνο στα γαλλικά και η συγγήτρια δεν ομιλεί την γαλλική. Οπότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Έπρεπε να μεταφραστεί η έκθεση για να μπορέσει ο εισηγητής να κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό μόλις τώρα καταλήξαμε να συζητάμε αυτό το θέμα, την Επιτροπή Αλίας και η παράταση του πρωτοκόλου λίγη τον Φεβρουάριο. Οπότε είμαστε στην τελευταία στιγμή πράγματι. Θα ήθελα να σας δώσω να σας πω τους δικούς μου λόγους για τους οποίους συνιστώ να μην συνενέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προσωρινή αυτή η παράταση του πρωτοκόλλου. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ πως είναι απαράδεκτο το Μαρόκο να παραμελεί εντελώς, να αγνοεί τα ερωτήματα της Κομισιόν για το όφελος θα έχει ο λαός της Δυτικής Σαχάρας. Δεν είπαν τίποτα από αυτού και θέλω να αναφέρω πως το 2009 η Επιτροπή Αλίας ζήτησε να επισκεφθεί το Μαρόκο για να μελετήσουμε βεβαίως κάποια στιγμή κάποια στιγμή το 2009 και το Μάιο λάβαμε μια επιστολή από την κυβέρνηση της αρχές του Μαρόκου που έλεγαν πως δυστυχώς ε, δεν μπορούσαν να μας δεχτούν ε, την περίοδο που ζητήσαμε. Η προτινόμενη περίοδος ήταν το 2010 ολόκληρο. Οπότε δεν ήθελα να πάμε δηλαδή απλούστοτα. Οπότε θεωρώ άρα πως το να συνενέσουμε σε αυτή τη συμφωνία ανταμείβει αυτές τις τακτικές του Μαρόκου που είναι εντελώς απαράδεκτες. Δεν απαντά, δεν δέχεται μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερον, εάν τώρα δείτε αυτή την μελέτη, η οποία υπάρχει και στα αγγλικά και στα γαλλικά, αν τη διαβάσετε, μιλάμε για την πιο αρνητική αξιολόγηση οποιασδήποτε αλληλευτικής συμφωνίας Πρώτα απ' όλα όταν μιλάμε για τα αποθέματα, τη βιολογική κατάσταση. Κατ' ουσίαν όλα τα αποθέματα είναι ε, υπεραλλιευμένα ή πλήρως αλλιευμένα πλην ε, ενός τη Ανδέλας στον νότο. Και αντιλαμβάνεστε πως ο νότος βεβαίως είναι τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Οπότε μόνο εάν αυξηθεί η εκμετάλλευση αυτού του αλλιεύματος ε, και βεβαίως μπορεί να πιάσει κανείς εκεί πέρα και σκουμπριά και στα σαυρίδια μαζί, στα δίχτυα, κάτι το οποίο είναι υπεραλλιευμένο ήδη και δεν θα το συνιστούσαμε. Πριν από λίγα λεπτά στην Επιτροπή Ελία είχαμε αυτή τη συζήτηση και κάποιο είπε «Μα ο στόλο τη Ευρωπαϊκής Ένωση αλλιεύει κλάσμα των αλλιευμάτων εκεί πέρα». Ε, ναι, αλλά παρόλα όλα αυτά. Είναι σημαντική η αρχή που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα πρέπει να έχουμε συμφωνίες μόνο εάν υπάρχει ε, κάποιο περίσσευμα από θέματος. Δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε τους ντόπιου ψαράδες. Και αυτό είναι λοιπόν ένα σημαντικό επιχείρημα για να απορρίψουμε αυτή την προσωρινή συμφωνία. Τρίτον, είναι η τομεακή στήριξη που βεβαίως αφορά την Επιτροπή μας. 13 εκατομμύρια 500.000 ευρώ το έτος είναι η στήριξη που θα έπρεπε να πάει για να στηριχθούν οι ντόπιοι αλληλείς του Μαρόκου. Η μελέτη της αξιολόγησης δείχνει πως μόνο ένα 15% του ποσού αυτού έχει χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει το λεγόμενο πρόβλημα απορρόφησης και το Μαρόκο δηλώνει πως το ποσό αυτό είναι μόνο 0,2% των συνολικών επενδύσεων στην αλληλεία του Μαρόκου. Στην περίοδο 2008-2010. Οπότε ο στόχος της αλληλευτικής πολιτικής του, πολιτικής του Μαρόκου να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή, οπότε η τομεακή στήριξη θεωρείται ασήμαντη για το Μαρόκο και οπωσδήποτε δεν έχει αναπτύξει τον αλληλευτικό τομέα στη χώρα αυτή. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της μελέτης αξιολόγησης, που επίσης δηλώνει πως έχει αποτύχει ε, αυτή η πολιτική και αυτό είναι βεβαίως σε μια οξία διατύπωση. Μία άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή της συμφωνίας είναι βεβαίως η κερδοφορία, η οικονομική πτυχή οι πλειοκτήτες της Ένωσης έχουν πληρώσει 1,9 εκατομμύρια ευρώ το έτος και 36 εκατομμύρια οι φορολογούμενοι. Οπότε 95% του κόστου συμφωνίας το πληρώνει ο δημόσιος τομέας. Μιλάμε για το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις αλληλευτικές μας συμφωνίες, αλλά ειδικά αυτή η συμφωνία ε, διαφέρει γιατί είναι και η λιγότερο αποτελεσματική ως προς το κόστος από όλες τις συμφωνίες. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, κάθε ευρώ που ξοδεύεται δημιουργεί 0,65 ευρώ προσθέμενης αξίας. Άμεσης και έμεσης προσθέμενης αξίας. Και πρόκειται για το χαμηλότερο λόγο κόστους προς όφελος από όλες τις παρόμοιες συμφωνίες. Επίσης, η συμφωνία αυτή δείχνει πως δεν έχει υπάρξει κάποια συμμόρφωση για την εκφόρτωση των αλλιευμάτων που έπρεπε να γίνεται στο Μαρόκο και επίσης αναφέρεται πως αυτό δεν σταθεροποιεί την ευρωπαϊκή αγορά καθώς μιλάμε για ένα οριακό ποσοστό των αναγκών της ευρωπαϊκής αγοράς. Επίσης, αναφέρω εδώ πέρα και την έκθεση αξιολόγησης, η οποία λέει πως αποτελέσματα είχαμε αλλά με πολύ υψηλό κόστος. Συνοψίζοντας, είχαμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού επίσης και η Επιτροπή Προϋπολογισμού επίσης συνιστά να μην συνενέσουμε στην ε, συμφωνία αυτή. Δεν είναι δηλαδή και από ε, οικονομική σκοπιά σωστή και ο εισηγητής της Επιτροπής Αλίας το ίδιο συνιστά να μην συνενέσουμε τη συμφωνία αυτή και η Επιτροπή ε, Ανάπτυξης επίσης και εγώ δηλαδή ο εισηγητής συνιστώ η Επιτροπή Ανάπτυξης να μην συνενέσει. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως ε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί λόγοι τους οποίους θα έπρεπε ίσως να γνωρίζαμε. Στο προηγούμενο Στρασβούργο θα ακούσατε πως ε, δεν ήθελε να στείλουμε το Κοινοβουλίο αυτή τη συμφωνία στο ελεγκτικό συνέδριο, κάτι το οποίο με απογοήτευσε, αλλά θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι θεωρούμε πως είναι σωστή ε, πλευρά. Ποιον πρέπει να ταχθούμε δηλαδή μετά την Αραβική Άνοιξη, εν πάση περιπτώσει. Και δεν πρέπει άρα να αγνοούμε το διεθνές δίκαιο, τις αρχές και τις περιβαλλοντικές ή ακόμα και τις οικονομικές. Οπότε προτείνω εν ολίγης να μην συνενέσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Madame Je passe à présent la parole Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τα μέλη. Ο κύριος Ντέβα θα πάρει πρώτος το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ πλήρως με την κυρία Λέβιν. Με μεγάλη υπομονή ανέφερε όλους τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Είναι εξωφρενική αυτή η κατάσταση. Η Σαχαράουι έχουν υποστεί επικισμό, μένουν σε στρατόπεδα και τους έχουν χτίσει και τείχος γύρω-γύρω, σαν το συνικό τείχος. Και εμείς κάνουμε τα στραβά μάτια. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Είτε αυτό το κοινοβούλιο και αυτή η ένωση έχει κάποιο νόημα ή δεν εκπροσωπεί τίποτα. Και αν εκπροσωπούμε κάτι, εκπροσωπούμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα προστασία του ασθενέστερου και το να ωφεληθούν οι φτωχότεροι και οι ασθενέστεροι. Ε, αυτοί είναι πραγματικά άνθρωποι ασθενέστεροι, τους έχουν περιορίσει σε στρατόπεδα εδώ και χρόνια. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση και δεν πρέπει να επιτρέψουμε τέτοια απεικιοκρατική συμπεριφορά. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να βοηθάμε και τις δύο χώρες και τις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε μια συμφωνία σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Οπότε, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πούμε φτάνει πια. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Monsieur Deval. La parole est maintenant à Monsieur Berman. Σας ευχαριστούμε, κύριος Μπέρμαν τώρα. Ευχαριστώ. Ε, εξ ονόματος του κ. Νόησερ του Σκιώδου, εισηγητή που δεν μπορούσε να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση, θα ήθελα να εκφράσω τον άκρατο θαυμασμό μου για αυτήν την τόσο συνοπτική πλην όμω σαφέστατη έκθεση που συνέταξε η κυρία Λέβιν. Είναι εξαιρετική ε, λόγω της επιχειρηματολογίας που εκεί παραθέτει, εξαιρετική επίσης ε, διότι έχει εκφραστεί με εξαιρετική ακρίβεια οι αλληλευτικές συμφωνίες, αυτή η αλληλευτική συμφωνία δεν επηρεάζει, ε, δεν έχει θετική ε, ε, επιρροή επί του κλάδου, ούτε και επί της απασχόλησης στο Μαρόκο. Πολύ λίγες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σχετικά με τις υποχρεωτικές ρήτρες εκφόρτωσης για τα νοσιακά αλληλεύματα. Δεν έχει γίνει τίποτα σεβαστό, δεν χρησιμοποιούνται χρηστά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ο λόγος του προς το όφελος είναι ιδιαίτερα χαμηλός και θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, ε, να εξετάσουμε δηλαδή με προσοχή τις επιμέρους διατάξεις της συμφωνίας για να ξέρουμε σε τι θα συνενέσουμε. Η νομιμότητα ε, της ε, συμφωνίας ε, είναι κάτι παραπάνω από αμφισβητήσιμη. Την περασμένη εβδομάδα όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς μεγάλη μου αγανάκτηση επέλεξε να μην ελέγξει την νομιμότητα της συμφωνίας. Σίγουρα όμως δεν υπάρχει θετική επιρροή. Καμία απόδειξη δεν υπάρχει ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην κατάσταση των Σαχράουι που βρίσκονται σε επισφαλέστατη θέση. Εάν λοιπόν δεν υπερασπιστούμε εμείς το κράτος το δικαίου, ποιος θα το κάνει κάνει. Ε, έχει την αμέριστη υποστήριξή μας η κυρία Λέβιν. Ευχαριστούμε. Ε, δίκαιο, έχετε καλά τα λέτε. Ο κύριος Βάιγκελ τώρα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συναδελφό μας και η συγγετρία, την κυρία Λέβιν, για την εξαιρετική της ε, παρουσίαση και να ευχαριστήσω και εσάς για το ότι πέρα από τη γνώση και τα δεδομένα το θέσατε το θέμα στο πραγματικό πολιτικό του πλαίσιο και σας συγχαίρω. Επίσης, αισθανθήκα πάρα πολύ άσχημα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο όταν είπαμε όχι στο διεθνές δίκαιο. Πρόκειται δηλαδή για δυσπιστία προς το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια συμπεριφορά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα το καλύτερο στον κόσμο για την ασφάλεια των μικρών κρατών και των φτωχών ανθρώπων από το διεθνές δίκαιο. Οπότε, πρόκειται για το εάν θα σεβαστούμε ή όχι το διεθνές δίκαιο και βεβαίως είναι πολύ πολιτικό το ζήτημα. Δεν θα μπω τώρα στην ε, καθαρά πολιτική πτυχή του προβλήματος, αλλά αρκεί να αναφέρω πως εδώ πέρα παίζουμε με την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εάν ακούσουμε μόνο τα συμφέροντα κάποιων χωρών και λόμπι κτλ. Έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου. Και το γεγονός πως το Μαρόκο συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε όταν ζητήσαμε δεδομένα για μια ξεκάθαρη εικόνα δηλαδή που θα πάνε τα λεφτά που σας δίνουμε για την αλληλεία μας δείχνει το πόσο ασφαλής θεωρούν εαυτούς ως δύναμη κατοχής σε μια περιοχή στην οποία δεν έχουν κανένα δικαίωμα να βρίσκονται. Η μόνη εντολή που έχει το Μαρόκο είναι να οργανώσει ένα δημοψήφισμα για την αυτοδιάθεση των Σαχαράουι και τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ε, απεικιοκρατία της, του χειρίστου είδους και είναι απαράδεκτη εντελώ. Οπότε για το λόγο αυτό και για τους λόγους που η συγγήτρια παρουσίασε σαφέστατα. Δεν νομίζω πως ε, έχουμε οποιαδήποτε άλλη επιλογή από το να πούμε όχι στη συμφωνία αυτή και να επιμείνουμε έναντι των εταίρων μας, το Μαρόκου δηλαδή εδώ πέρα, ε, θα πω μόνο το εξής. Όταν συζητούσαμε τελευταία φορά τη συμφωνία αυτή, και η στάση μας και η πρόταση του συναδέλφου του κυρίου Νταφ ε, για το εάν θα πάμε στο 10 ή όχι κρινόταν πολλοί συνάδελφοι έλεγαν να, λάβουμε υπόψη ε, το ότι το Μαρόκο είναι αυτό που λέμε η μόνη δημοκρατική χώρα αυτή τη στιγμή ε, μεταξύ των αραβικών χωρών. Ένας λόγος παραπάνω για να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το επιχείρημα για να ε, κάνουμε εκπτώσεις στην παράνομη συμπεριφορά. Οπότε η μόνη σωστή θέση είναι να μην στηρίξουμε τη συμφωνία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πόγκα τώρα. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της ε, και ίσως τώρα θα πάω ενάντια στο ρεύμα όλων αυτών των δηλώσεων που έχουμε ακούσει ε, στη σημερινή μας συζήτηση. Όντως θα σας πω ότι δεν συμμερίζομαι την άποψη της εισηγήτριας. Είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου η Επιτροπή μας ε, να ταχθεί υπέρ της έγκρισης για δύο λόγους. Πρώτον, για ένα Τεχνική φύση λόγω. Πρόκειται για μια προσωρινή συμφωνία που εφαρμόζεται ήδη από το Φεβρουάριο του 2011 και που εκπνέει το Φεβρουάριο του 2012. Οπότε στην πράξη το συμφέρον της απόρριψης είναι μηδαμινό σε σχέση με την κατάσταση των αλλιευμάτων. Έχουν ήδη αλλιευθεί, έχουν ήδη πολυθεί τα ψάρια. Δεν μπορούμε πλέον να τα επιστρέψουμε εμείς στη θάλασσα, στον υδάτινο βίο τους. Τώρα για την, κλαδική διάσταση, αν θέλετε, του πρωτοκόλου, του, του τομέα της αλλίας, ε, Ε, θα, εδώ θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο το να αναθεωρήσουμε την ε, τομεακή αυτή βοήθεια που χορηγείται στο Μαρόκο. Δηλαδή θα έπρεπε να ε, αποζημιώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μαρόκο ένα κομμάτι της βοήθειας που ήδη έχει χορηγηθεί ε, στον τομέα της Αλίας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει, υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της έγκρισης συμφωνίας. Εξελίσσεται το Μαρόκο, υπάρχει ένας μεταρρυθμιστικός που πνέει και στο Μαρόκο μετά την Αραβική Άνοιξη και άρα είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτή τη χώρα στι μεταρρυθμίσει που έχει αναλάβει και να στείλουμε ένα σήμα ανοίγματο, διαλόγου. Η απόρριψη δεν θα γίνει κατανοητή κατά τη γνώμη μου από τον ντόπιο πληθυσμό γιατί μα γυρίζει την πλάτη τη η Ευρώπη ενώ κάνουμε μεταρρυθμίσει ε, στον τομέα τη διακυβέρνηση, θα αναρωτηθούν όλοι οπότε Πρόεδρε ε, θα υποβάλω σύντομα μια τροπολογία που θα καλεί το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη συμφωνία. ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπέγμα ε, μου ζήτησε το λόγο. Κύριε Πόγκα, μία διευκρίνηση. Όταν λέτε, όταν διαβάζετε την έκθεση του Καρλ Χάγκλουντ, θα ε, καταλαβαίνετε ε, πέραν κάθε αμφιβολία, σε γιατί σημειώθηκε αυτή η καθυστέρηση ως προς την εξέταση από πλευράς του Κοινοβουλίου της Αλληλευτικής Συμφωνίας. Αυτό που έγινε είναι ότι αναπέμφθηκε η έκθεση στο Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2011, ενώ ήδη ήταν σε ισχύ από το Φεβρουάριο, όπως σωστά είπατε. Ε, πρόκειται για ένα σφάλμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ουχή του Κοινοβουλίου, άρα δεν θα έπρεπε εμείς να σταματήσουμε τώρα να ασκούμε ε, πλήρως τα δημοκρατικά μας δικαιώματα λόγω ενός σφάλματος της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, με διευκολύνει πολύ η παρέμβαση του κυρίου Πόγκα, διότι ουσιαστικά όλα αυτά που είπε ε, συμπίπτουν ε, με τη δική μου στάση. Τι συμβαίνει εδώ, υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που μπερδεύουμε, που αναμειγνύουμε και υπάρχουν και κάποια πράγματα που λέγονται και δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Λέγεται ότι υπάρχουν παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί Υπάρχουν επιστοποιήσεις με απόλυτα έχει και στο επίπεδο του Ηνωμένων Εθνών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σχέση με την διεθνή νομιμότητα. Πράγματι υπάρχουν όλα αυτά. Εγώ ε, αυτό που μπορώ να σας πω εδώ είναι ότι πράγματι η διεθνής αυτή συμφωνία δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Ε, ο λόγος μου έχει την αξία που έχει. Ε, και είναι σίγουρα το ίδιο σοβαρός με αυτούς που λένε ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να αναφερόμαστε σε ξένους φορείς που θα πιστοποιήσουν δεν θα πιστοποιήσουν, αφού έχουμε τα πιστοποιητικά. Τα έχουμε εδώ. Άρα υπάρχει ένα πολιτικό θέμα, πολύπλοκο πολιτικό θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Και κάποιοι από τους παρόντες, κάποιες από τις πολιτικές ομάδες που εκπροσωπούνται εδώ ίσως, με τα λόγια μπορεί να ήταν λίγο πιο επιθετικές, επιθετικής ό,τι αφορά την αλληλεγγύη με τους ε, Σαχαράου. Εγώ πραγματικά συγκινήθηκα όταν άκουσα τον κύριο Ντέβα να μιλά για την ευθύνη, για τους ε, καταβλισμούς, τους μη καταβλισμούς. Μα πού είναι οι καταβλισμοί, αυτό δεν μας είπε ο κύριος Ντέβα όμως. Οι καταβλισμοί στους οποίους αναφέρθηκε ο κύριος Ντέβα. Πού βρίσκονται, σε έδαφος ποιου κρατού, κράτους υπάρχει, ποια δύναμη έχει αυτά τα στρατόπεδα, αυτούς τους καταβλισμούς ε, στο έδαφος της και πώς και ποιοι τα διαχειρίζονται, υπό ποια ε, γίδα βρίσκονται κάτω από ποια αρχή βρίσκονται, την εποπτεία τους, ποιος την έχει και το ότι αυτή τη στιγμή παραμένουν και επιβιώνουν αυτά, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά τα στρατόπεδα, για αυτούς τους καταβλισμούς. Ποιος συμβάλλει στο να υπάρχει υγεία και παιδεία υπ' αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες σε αυτούς τους καταβλισμούς που δεν είναι στο έδαφος ούτε της Σαχάρας ούτε του Μαρόκου, ε. Δεν πρέπει να τα έχουμε και αυτά υπόψη μας, εκτός εάν θέλουμε να τα γνωρούμε ή αν τα γνωρούμε απλά. Λέτε, ποιες θα ήταν επιπτώσεις από μια αναστολή, κάτι που δεν είναι συμφωνία, αλλά είναι παράταση μια συμφωνίας που έχει ήδη παραταθεί, ώστε να είναι δυνατό να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συμφωνία. Υπήρξε μια συμφωνία, παρατάθηκε η συμφωνία αυτή, υπό την προϋπόθεση θα διαπραγματευτούμε στη συνέχεια μια καλύτερη συμφωνία. Λοιπόν, λίγη τον Φεβρουάριο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα και από το Φεβρουάριο ή μέχρι το Φεβρουάριο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία που θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο, θα συνάδει με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνάδει και με τα συμφέροντα του Μαρόκου. Και βέβαια από αυτή τη συμφωνία θα ωφελείται ο πληθυσμός του εδάφου στα έδω του οποίου θα ε, γίνεται η αλίευση. Αυτή είναι η όρη θέλουμε να διαπραγματευτούμε μια καλύτερη συμφωνία σε όλους αυτούς τους τομείς, που θα είναι πιο ευεργετική συμφωνία για το Μαρόκο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια κυρίως για τον πληθυσμό, στα ύδατα του οποίου θα μπορεί κανείς να αλλιεύει. Αυτό είναι το ερώτημα, αυτό πρέπει να σας απασχολήσει. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις. Πολύ καλά. Το είπε ο κ. Ε, Πογκάν και συντόμως. Αν ανασταλεί η παράταση κάτι που ήδη λειτουργεί επί 7 μήνες και που απομένουν 4-5 για να λήξει. Ποια θα είναι οι επιπτώσεις της αναστολής ισχύω. Τούτου λεχθέντος, και ως μέλος Επιτροπής συμφωνώ με αυτό που ο κύριος Πόγκα, ακούστε, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι, βάσει της εμπειρίας που έχουμε με άλλες χώρες. Έχω την εντύπωση ότι το Μαρόκο δεν ενδιαφέρεται και τόσο να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Και αν το Μαρόκο δεν ενδιαφέρεται και τόσο, ας το αφήσουμε το Μαρόκο. Πρέπει να δούμε ποια είναι η εναλλακτική. Το Μαρόκο και άλλες τόσες αφρικανικές χώρες, τι εναλλακτική λύση πρότειναν ή θα προτείνω να του πούμε ότι δεν πρόκειται να επιμηκύνουμε, να παρατείνουμε, να επαναπεβεβαιώσουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν ξέρετε ε, ότι υπάρχουν και άλλοι συνομιλητές. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Υπάρχει μια χώρα μήπως που λέγεται Κίνα, που λέγεται Ιαπωνία, που λέγεται Ρωσία, που, λέγεται, που υπογράφουν αυτές οι χώρες ε, συμφωνίες με το Μαρόκο που δεν ε, θέλει να υπογράψει. Sorry λέτε κύριε Ντέβα, όχι sorry. Φυσικά και δεν συμφωνείς. Δεν συμφωνείς τόσο που ούτε και εγώ συμφωνώ. Ε, εντάξει, δεν συμφωνούμε. Δεν... Μπορούμε να μην συμφωνούμε. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε ουσιαστικά. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα. Νομίζω ότι το Μαρόκο σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, δεν πολύ ενδιαφέρεται. Και μου δίνει την εντύπωση ότι η συμφωνία που εντέχεται να ε, διαπραγματευτούμε, για την αλληλευτική συμφωνία με το Μαρόκο μιλάω, που μακάρι να είναι μια καλύτερη συμφωνία σε κάθε επίπεδο να είναι πιο ευεργετική για το Μαρόκο, να εκπαιδεύτούν καλύτερα οι αλληλείς, να ζήσουν καλύτερα αυτοί που ζουν στη Σαχάρα. Αυτοί που ζουν στη Σαχάρα, έτσι ε, το ξαναλέω, ο πληθυσμός που ζει στη Σαχάρα να ωφεληθεί. Όχι κάποια πολιτικά ε, καθεστώτα ή δομές που δεν ζουν στη Σαχάρα όμως. Εγώ νομίζω ότι το Μαρόκο μπορεί να ενδιαφέρεται για την διαπραγμάτευση μιας άλλης αληθικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο θα ενταχθεί σε άλλη σειρά συμφωνιών που ενδέχεται να ενδιαφέρουν πολιτικά και οικονομικά το Μαρόκο. Αυτή Αλλιώ σε θέματα αλλιώ το Μαρόκο έχει άλλου συνομιλητέ οι οποίοι περιμένουν έχουν στηθεί στην ουρά και περιμένουν να ε, συμφωνήσουν, να υπογράψουν συμφωνία με το Μαρόκο, πολύ πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι αυτή που υπογράψαμε εμεί με το Μαρόκο. Άρα θα είναι πολύ πιο σοβαρές και οι επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών για την Αλία. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν κάνουμε μια σύγκριση με τη Σενεγάλη, που εντάξει εκεί η Αλία δεν είναι, γίνεται όπως γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι σέβονται τα είδη, τα αλλιευτικά κτλ. Γιατί αυτοί υπογράφουν συμφωνίες με χώρες από τις οποίες εμείς έχουμε εξαφανιστεί. Και έπονται άλλοι έπονται άλλοι και αυτοί δημιουργούν, αυτοί που υπογράφουν συμφωνίες εκεί που εμείς δεν έχουμε υπογράψει, αυτοί λοιπόν δημιουργούν ε, μεγάλο πρόβλημα και καταστρέφουν την αλία. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε, δεν θα ψηφίσουμε, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι σχετική η σημασία αυτού. Μιλάμε για τέσσερις μήνες ε, ουσιαστικά, έτσι. Και αν μέσα σε αυτού του τέσσερι μήνε ή μετά δεν καταφέρουμε να επαναδιαπραγματευτούμε μια σοβαρή αποτελεσματική ενδιαφέρουσα συμφωνία που να μα φαίνεται σε όλου θετική, δεν πάμε πουθενά. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το μόνο για το οποίο πρόκειται εδώ είναι μια μικρή, πολύ σχετική κίνηση, μια πολύ σχετική χειρονομία. Και συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πόγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαρτίνες. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Αλεξανδρό από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να είστε και σύντομος. Oui. Merci, madame. Je vais essayer Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Αλλά ο αριθμός των παρεμβάσεων καταδεικνύει και το ενδιαφέρον που δείχνει η Επιτροπή σας για αυτό το φάκελο που είναι κατεξοχήν συμβολικός και σημαντικός. Θα περιοριστώ στα πλέον ουσιαστικά στοιχεία και εγώ μόλις τώρα ήρθα από τη συνεδρία της Επιτροπής Αλίας όπου ήταν η συγκεντριά σας και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις διάφορες ε, ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να ρίξω ένα νέο φως επίσης ε, στην ε, συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα την κυρία Λέβιν. Συνέταξε μια πάρα πολύ καλή έκθεση παρά τις διαστάσεις απόψεων που μπορεί να σημειώνονται για επιμέρους σημεία. Επίσης, κατά την παρουσίαση, ε, με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, παρέθεσε όλη της, ε, την επιχειρηματολογία και την υποστήριξε με συγκεκριμένα στοιχεία όπως το συνηθίζει. Συγχαρητήρια λοιπόν και υπάρχουν στοιχεία που αξίζουν να μας προβληματίσουν. Ε, αξίζει να μας προβληματίσουν. Ε, Καταρχήν θα ήθελα να σχολιάσω την καθυστέρηση που σημειώθηκε στη διοικητική διαδικασία στα διάφορα θεσμικά όργανα και κατόπιν να σχολιάσω την ε, υπογραφή του πρωτοκόλλου που έγινε, αν θυμάμαι καλά, στις 27 Φεβρουαρίου του 2011. Λυπούμεθα για την καθυστέρηση που ε, σημειώθηκε. Ο εισηγητής της Επιτροπής Αλίας επίσης Λυπάται διότι η έκθεση αξιολόγηση ε, είναι σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνει. Καταλαβαίνουμε την απαγοήτευσή του, ε, τη δυσαρέσκειά του και ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταφραστεί η έκθεση αξιολόγησης σε μια γλώσσα που να κατανοεί ούτως ώστε να κατανοήσει όλα, όλες τις λεπτές χρειές αν θέλετε του ζήτηματος. Έγινε λοιπόν η μετάφραση. Η έκθεση αξιολόγηση ε, έγινε από εξωτερικό σύμβουλο και αληθεύει ότι η έκθεση αυτή ε, δεν ε, είναι ουδόλως ικανοποιητική. Αληθεύει επίσης ότι είναι λίγο παλιά η έκθεση αυτή και έκτοτε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μιλάμε για απορρόφηση από πλευρά των μαροκινών αρχών κονδυλίων που κανονικά θα διοχετεύονταν στην τομιακή βοήθεια. Πριν από αυτό το πρωτόκολλο αληθεύει και είχαμε δηλώσει τη δυσαρέσκειά μας και το είχαμε τονίσει επανελειμμένα σε επαφές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές. Αληθεύει λοιπόν ότι είχε σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση, άρα κακή απορρόφηση των κονδυλίων. Οι Μαροκινοί επικαλέστηκαν μία σειρά λόγων, ανέμεναν την εκπόνηση της εθνικής αλλιευτικής τους πολιτικής και μετά την ε, έγκριση και την ε, εφαρμογή αυτής της πολιτικής διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό απορρόφηση ε, των κονδυλίων σαφέστατα βελτιώθηκε στο ενδιάμεσο διάστημα, όμως εκπονήθηκε αυτή η έκθεση αξιολόγηση και αυτή η μικρή βελτίωση ε, δεν εκάλυψε το κενό. Πρόκειται για λεπτομέρεια βεβαίως, αλλά καλό είναι να τονίσουμε. Διάφορα μέλη της Επιτροπής σας αναφέρθηκαν στην κατάσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων του Μαρόκου. Εάν διαβάσει κανείς με λίγαν αντικειμενικό τρόπο και με ακρίβεια το περιεχόμενο της έκδοσης αξιολόγησης ε, φαίνεται ότι ο η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται εκεί για όλα τα ελευτικά αποθέματα είναι κάτι αναμφισβήτητο. Όμως το πρωτόκολλο καλύπτει πολύ περιορισμένο αριθμό αποθεμάτων συγκεκριμένα καλύπτει αλλιεύματα αεραστεχνικής αλληλείας από πλευρά Σιβηρικής ε, Χερσονήσου και ε, καλύπτει και κάποια πελαγικά, πελαγικά είδη. Ε, ε καλύπτει τα, δεν καλύπτει η συμφωνία τα καρκινοειδή. Δεν καλύπτει λοιπόν τα οστρακοειδή μετά από διαπραγμάτευση με τις ε, μαροκινές αρχές, ε, διότι ήταν σε τέτοια κατάσταση το ελευτικό απόθεμα που δεν ήταν ε, δυνατό να συνεχίσουμε να το απομιζούμε. Για, ως προς τα αποθέματα λοιπόν, είναι πολύ γενική η εικόνα που δίνεται μέσα στην έκθεση, ενώ οι πληροφορίες θα έπρεπε να περιορίζονται στα αποθέματα που όντως καλύπτονται από το εν λόγω πρωτόκολλο. Ε, σχετικά με τη φύση του πρωτοκόλλου τώρα, πρόκειται για διάρκεια 12 μήνη και γιατί το διαπραγματευτήκαμε αυτό το πρωτόκολλο, διότι θέλαμε να έχουμε τις περισσότερες νέες πληροφορίες ε, ή δυνατόν πληροφορίες, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει ή όχι μια πραγματική διαπραγμάτευση για ένα μελλοντικό πρωτόκολλο. Το μελλοντικό πρωτόκολλο εξορισμού θα έχει πολύ ανώτερη διάρκεια σε σχέση με τους 12 μήνες που ισχύουν για το τωρινό. Αυτό το πρωτόκολλο, το μονοετές, συνιστά μια παρένθεση, ένα διάμεσο στάδιο, αν θέλετε, και είναι πρόδρομος μιας ε, ε, δυνάμει διαπραγμάτευσης για τη σύναψη νέου αλευτικού πρωτοκόλλου. Έχετε άλλο ένα λεπτό γιατί ήδη μιλήσατε πέντε λεπτά και έχουμε και μεγάλη καθυστέρηση. Ε, εντάξει, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, αλλά είχα διάφορα μηνύματα που ήθελα να περάσω ε, στους ακροατές και θεωρούσα ότι είναι καθήκον μου να το κάνω. Λοιπόν, δεν έγινε πραγματική διαπραγμάτευση για αυτό το πρωτόκολλο, διότι το πρωτόκολλο επαναλαμβάνει αυτούσεις ε, τις διατάξεις ε, του προηγουμένου, με μία σημαντική βέβαια εξαίρεση, δηλαδή υποχρέωση υποβολής έκθεσης αναφοράς από πλευράς των Μαροκινών Αρχών σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πρωτόκολλο επί το σύνολο των διοικητικών περιφερειών του Μαρόκου. Καλύψαμε δηλαδή και την γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων, κάτι που απουσίαζε από το προηγούμενο πρωτόκολλο. Αυτό είναι στα προσθέμενη αξία σε σχέση με το προηγούμενο, η οποία θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε πρώτες εκπνοίες του πρωτοκόλλου, το κατά το κατά πόσο θα πρέπει να ξεκινήσουν πραγματικέ διαπραγματεύσει με τι μαροκινές αρχέ για τη σύναψη ενός νέου πρωτοκόλλου. Νομίζω ολοκλήρωσε και, και κυρία Πρόεδρε, νομίζω δεν μπορείτε παρά να δηλώσετε ικανοποιημένοι, διότι δεν υπερεύει το χρόνο μου. Βεβαίω, όπω και όλοι οι υπόλοιποι, λέει η Πρόεδρο, Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Λέβιν ε, για τα συμπεράσματα τη συζήτηση Και κυρία Λέβιν, μην ξεχαστείτε και εσεί σύντομα. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος ε, Πόγκα. Είπε πως εάν δεν εκρίνουμε τη σημασία, τι σημασία έχει, δεν μπορούμε να ξαναρίξουμε τα ψάρια στο νερό. Όχι, όχι. Πράγματι αυτό ισχύει, αλλά όπως επεσήμανε και ο κύριος Μπέρμαν, πρόκειται για την πρώτη δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο για να εκφέρει άποψη επί της συμφωνίας αυτής. Ε, δεν φταίμε εμείς λοιπόν, άρα και η αρχή είναι εξίσου σημαντική επίσης. Οπότε, εάν μιλάμε για υπεραλληλία ε, ή για οτιδήποτε άλλο, δεν έχει σημασία. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ε, αποζημιώσουμε βεβαίως το Μαρόκο για τους 8 μήνες αυτούς αλίας. Επίσης, για την κατάσταση για τον κλάδο Εάν ε, δεν συμφωνήσουμε σε αυτή την συμφωνία θα παρατηρήσουμε σύντομα στην Επιτροπή Ελίας και στην Επιτροπή μας που θέλει να πάει το Κοινοβουλίο ε, αλλά έχουμε και ψηφοφορία στην Ολομέλεια οπότε θα έχει χρόνο ο Ευρωπαϊκός Κλάδος Αλίας να προσαρμοστεί. Οπότε θα ήθελα να τονίσω και πάλι πως δεν είχαμε συμφωνία μεταξύ 99 και 2007 και τα κατάφερε ο ευρωπαϊκός κλάδος της αλίας, δεν υπήρχε πρόβλημα. Οπότε δεν είναι το τέλο του κόσμου. Όταν μιλάμε τώρα για την τομεακή στήριξη, εγώ συνάντησα την Επίτροπο πριν από λίγες εβδομάδες, δεν υπήρχε τότε μια νέα αξιολόγηση για το πώς ε, έχει εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία στο Μαρόκο. Βεβαίω μπορεί να έχει υπάρξει κάποια βελτίωση στη λεγόμενη δυνατότητα απορρόφησης του Μαρόκου η οποία ήταν πάρα πολύ χαμηλή πέρσι. Η Επιτροπή δεν πλήρωσε καν ε, το πλήρες ποσό τομεακής στήριξης γιατί δεν είχε χρησιμοποιήσει με το σωστό τρόπο τα κονδύλια το Μαρόκο. Οπότε η αναπτυξιακή πτυχή της συμφωνίας αυτής δεν ε, έχει ληφθεί υπόψη. Το Μαρόκο επενδύει το ίδιο στον τομέα της Ελίας και δεν έχει χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια και θεωρώ πως μια νέα συμφωνία με το Μαρόκο είναι, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξέταση, αλλά βεβαίως θα έπρεπε να αφορά μόνο τον Βορρά και αυτό ακριβώς πρότεινε η Επιτροπός Αλίας. Ήθελε μία εντολή να πάει να διαπραγματευτεί μόνο για τον Βορρά, αποκλείοντας δηλαδή την Δυτική Σαχάρα. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Και στον κύριο Μαρτίνες θα έλεγα πως αυτό θα διευκόλυνε και τον ε, ισπανικό αλλιευτικό κλάδο που αλλιεύει σε γειτονικά νερά. Πρέπει να έχουμε κάποια συμφωνία για να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα, αλλά όχι με τα ύδατα της Δυτικής ε, Σαχάρας. Και δυστυχώς αυτό δεν το δέχτηκε τότε η Κομισιόν, αυτό ήταν πριν από τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, αλλά θα ήθελα να τονίσω πως πάρα πολλά κράτη-μέλη καταψήφισαν τη συμφωνία αυτή στο ε, Συμβούλιο, οπότε δεν είναι και ένα θέμα δηλαδή στο οποίο συμφωνούν όλοι. Πρέπει λοιπόν να το λάβουμε αυτό πάρα πολύ σοβαρά υπόψη στην Επιτροπή μας και στο Κοινοβούλιο πριν ε, αρχίσουμε να δικαιολογούμε μια συμφωνία η οποία μπορεί σε ένα έτος να μας φαίνεται πως μας εκθέτει εάν ε, πούμε ναι στην αλία σε κατεχόμενες περιοχές. Όπως ντρέπονται τώρα κάποιες χώρες για τις σχέσεις τους με την Ισία, Αίγυπτο, Λιβύη κτλ. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών για αυτό το σχέδιο έκθεσης εκπνέει στις 17 Οκτωβρίου ακριβώς στις 12 το μεσημέρι να βάλω και τα γυαλιά μου. Οι συντονιστέ τη Επιτροπή Ανάπτυξη, όπω ξέρετε, πήραν την απόφαση να προσκαλέσουν μετά από αίτηση του κυρίου Λουί Μισελ, τον κύριο Ρόμπ Βόσα, είναι συντονιστή τη ομάδα προβληματισμού σχετικά με την καθυστέρηση που σημειώνεται ω προ την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία για την ανάπτυξη. Ε, ε, θεσπίστηκε αυτή η ομάδα από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια ομάδα προβληματισμού και συναποτελείται από 20 επιμέρους οργανισμούς περίπου των ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, καθώς και η ο, ο, ο, ο ΑΣΑ και ο Επίσης η ομάδα ε, παρακολουθεί την υλοποίηση του 8ου στόχου της ε, χιλιετίας, ε, δηλαδή μια παγκόσμια αναπτυξιακή εταιρική σχέση, εντατικοποιώντας τον, την οργανική συνεργασία. Κύριε Βός, συνειδητοποιούμε ότι η εταιρική σχέση είχε βασικά επιτεύγματα με ένα ύψος ρεκόρ της αναπτυξιακής βοήθειας για το 2010, κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αλλά επειδή πλησιάζει το 2015 αυτός ο αργός ρυθμός υλοποίησης και το εύρος της πρόοδου που αναμένεται να σημειωθεί καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να δραστηριοποιηθούμε. Υπάρχουν σημαντικότατες προκλήσεις για τις παγκόσμιες δωρητές ΕΔΕ λόγω των διεθνών εξελίξεων. Κύριε Βός, θα σας δώσω το λόγο και ευελπιστώ να είναι καρποφόρα η ανταλλαγή απόψεων εκεί για σας και για μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ε, thank Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Σας παρουσιάσω την έκθεση που ανέφερε πέρας. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα προσπάσω να είμαι σύντομος. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και μια συζήτηση πάνω στο θέμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω, όπως είπε και η Πρόεδρος, ε, είναι η ειδική αυτή έκθεση της ε, Task Force ε, για το 2011 και το 2010, ενημερωμένη, επικαιροποιημένη λοιπόν έκθεση. Και ένα από τα βασικά μηνύματα αυτής της έκθεσης είναι να δούμε τι γίνεται μετά από τη Σύνοδο Κορυφής του 2010 για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας Πώς έχει κατάσταση λοιπόν, έχουμε διάφορα έγγραφα στα οποία αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχουμε επιτύχει προς την επίτευξη των στόχων αυτών, αλλά σίγουρα για πολλούς στόχους δεν έχουμε σημειώσει την απαντούμενη πρόοδο και φοβόμαστε ότι πολλές χώρες ίσως να μην καταφέρουν να τους πετύχουν εγκαίρως αυτούς τους στόχους. Το ίδιο ισχύει και για διάφορα μέρη της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, όπου δεν έχουν ε, τηρηθεί όλες οι αναλυφθεί σε δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Επανεπιβεβαιώνουμε και προσθέτουμε κάποιες δεσμεύσεις. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεκτικότητα με άλλους τομείς και άλλες ατζέντε, βιώσιμη ανάπτυξη για παράδειγμα, βοήθεια, εμπορική βοήθεια και ανακούφιση του χρέους και άλλους τομείς. Ταυτόχρονα θέλουμε να είναι τέτοια αυτή η συνεκτικότητα ώστε επιτυχείς πολιτικές στις ανεψόμενες χώρες να αναβαθμιστούν ε, ακόμη περισσότερο ώστε να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στις προσπάθειες των ίδιων των χωρών για μεγαλύτερη ιδιοκτησία, εθνική και οικειοποίηση των όλων διαδικασιών, να ενισχύσουν ε, τις πολιτικές που οι ίδιες θα αποφασίσουν και βέβαια θέλουμε να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες εταιρικέ σχέσεις και να τηρήσουμε τις μέσες που έχουμε αναλάβει, αλλά αυτές οι ε, προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο να ευθυγραμμιστούν με αυτές τις εταιρικές σχέσεις. Στο τέλος θα αναφέρω και το ότι ζητήσαμε από την γραμματεία του ΟΗΕ να αρχίσει να εξετάζει το περίγραμμα μιας ε, ε, ατζέντας για μετά το 2015 που είναι και ο στόχος για να έχουμε πληρώσει τους στόχους, τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας όπως γνωρίζετε. Άρα μας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να σας δώσω όλα τα μηνύματα της έκθεσης βέβαια, θα ήθελα να τονίσω πάντως κάποια από αυτά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια αίσθηση κατεπήγοντο. σίγουρα μεν ισχύει ο στόχος του 2015, σε ό,τι αφορά τις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις που θα πρέπει να στηρίξουν ε, τις εθνικές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε το 2015 για να ε, εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι. Αν υπάρχει στήριξη μέσω των εθνικών προσπαθειών μπορούμε να επιταχύνουμε το ρυθμό. Υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του κατεπήγοντος. Επίσης υπάρχουν κάποιες ε, ημερομηνίες λήξεις ε, όπως παραδείγματο χάρη δεσμεύσεις σε Glen οι οποίες ήδη έχουν λήξει. Έπρεπε κάποιοι στόχοι να είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2010. Έχουμε και το HIPIC, το μηχανισμό ανακούπησης κρέου ε, που ε, παρότι έχει λήξει από το 2006 συνεχίζει μεν, αλλά ο μηχανισμός δεν μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή νέων χωρών ή να ε, παράσχει περισσότερη ανακούφιση από το χρέος σε χώρε που αντιμετωπίζουν ακόμη προβλήματα. Μια άλλη ανησυχία είναι ότι σε παγκόσμιε εταιρικέ σχέσει υπήρξε κάποια πρόοδο, αλλά όχι αυτοί που είχε, είχαν υποσχεθεί οι χώρες ε, στην διάρκεια της διάσκεψης κορυφής. Δεν θα επισέλθω σε όλα τα ζητήματα, θα σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα στον τομέα της βοήθειας και του εμπορίου. Ίσως γνωρίζετε τα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι καλό είναι κάποια από αυτά τα θέματα να τα επισημάνω. Ξέρετε ότι οι στόχοι Glen Eagles από την ε, ομάδα των 8 στην πόλη αυτή της Σκοτίας πρώτο ε, αναφέρθηκαν και ορίστηκαν αύξηση 2010 ε, για τη βοήθεια και μάλιστα για την περίπτωση Αφρικής διπλασιασμού της βοήθειας. Ναι, μεν έχουμε σημεία ρεκόρ στην αύξηση της βοήθειας σε απόλυτους όρους, αλλά ε, υπολοιπόμεθα κατά 21 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τους στόχους Glen Eagles και για την Αφρική ναι μεν αυξήθηκε η βοήθειά μας αλλά πάλι υπολείπεται κατά 18 δις επίσημα και βοήθεια για την Αφρική. Άρα δεν τηρήθηκαν οι στόχοι ε, και οι δεσμεύσεις Glen Eagles. Έχουμε λοιπόν άλλους άμεσους στόχους ε, για μετά το 2010 ναι, μεν αυξήθηκε η βοήθεια και ε, εν καιρό ύφεση, αλλά για τις ε, προβλέψεις μας βλέπουμε ότι θα παραμείνει σε τέλμα η βοήθεια, άντε το πολύ να αυξηθεί κατά 1% την επόμενη τριετία, που σημαίνει ότι και μετά την ημερομηνία λήξη του οι στόχοι Glenn English δεν θα επιτευχθούν. Τώρα, στόχο των Ηνωμένων Εθνών ε, πολλέ φορέ σε πολλά βήματα συζήτηση επανεπιβεβαιώνεται και στην ε, Σύνοδο Κορυφή για τους Αναπτυξιακούς στόχου Ηλιετία και σε άλλες ε, διασκέψεις ε, μιλάμε για αυτό το στόχο του 0,7% αλλά μόνο πέντε χώρες έχουν επιτύχει το στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχουμε θέσει ως στόχο το 2010 να φτάσουμε στο 0,51% του Εθνικού Ακαθάριστου Εισοδήματος των Δωρητών στόχος που δεν έχει επιτευχθεί εξ ολοκλήρου. Έχουμε δηλαδή κάνει λίγο παραπάνω από το μισό για να φτάσουμε στο ε, μεσόρο. Αν λοιπόν θέλει η κοινότητα των δωρητών να τηρήσει τις δεσμεύσεις και υποσχέσεις που έχει αναλάβει, θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα τα επόμενα χρόνια και παρά την κρίση, παρά την ύφεση. Και ο Γενικός ε, Διευθυντής, το αφεντικό μου, λέει ότι πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε η ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση και η κρίση να αποβεί ε, σε βάρος των φτωχών και των ευάλωτων ε, που χρειάζονται αυτή ε, τη βοήθεια. Πρέπει λοιπόν να γίνουν επενδύσεις στο μέλλον για όλον το όφελος. Στην έκθεσή μας επίσης τονίζουμε το θέμα της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, όχι μόνο του μεγέθους της βοήθειας. Υπάρχουν πολλά αναλυτικά στοιχεία, αλλά εγώ θα επιμείνω σε τρία μόνο. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε τη δήλωση των Παρισίων για την ανάγκη αποτελεσμα... μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας έχουμε ε, πίνακε πίνακες ε, βαθμολογίας, πίνακες επιδόσεων και μάλιστα πριν από 10 ημέρες δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία και μας δίνουν μια αρκετά ε, ζωφερή εικόνα. Ένας από τους στόχους μόνο ε, από τους 13 έχουν επιτευχθεί, 12 δηλαδή δεν τους πετύχαμε και νομίζω ότι το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι πρώτον η πρόοδος που σημειώθηκε η σημαντικότερη είναι από τις αποδέκτριες χώρες που κατάφεραν να βελτιώσουν ε, και να διατυπώσουν εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους με τους οποίους μπορούμε να συμφωνήσουμε ως επιτοπλίστων, αλλά αυτό το οποίο υποσχέθηκε η κοινότητα των δωρητών, δηλαδή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οι περισσότερες ε, υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν. Υπήρξε εκπρόοδος σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά αν βλέπουμε ότι οι 12 από τους 13 στόχους δεν τηρούνται, αυτό σίγουρα ε, δεν εμπνέει και μεγάλη ισοδοξία, δημιουργεί ανησυχία. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, είναι δύσκολη πρόοδος σε αμψόμενες χώρες, δεν ξέρουμε την εξωτερική χρηματοδότηση που μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάθε χρόνο για τις χώρες αυτές, άρα και αυτές οι χώρες δυσκολεύονται και για την ε, απόδοση της βοήθειας υπάρχουν ε, στόχοι, υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι δείκτες και αυτό μπορεί να γίνει με διμερή ταμεία ή με εγκάρσια, με διμερή ενισχύση ή με εγκάρσια ταμεία. Αυτές λοιπόν είναι οι ανησυχίες μας γιατί δεν έχει το πρόβλημα να κάνει μόνο με το μέγεθος της βοήθειας αλλά και με την αποτελεσματικότητα και τη συνεκτικότητα δηλαδή πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η βοήθεια ε, εφαρμόζεται για και συνεργάζεται με τι εθνικέ αναπτυξιακέ πολιτικέ και στρατηγικέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ίδιε τι δεσμεύσει, οι δωρητέ αναλαμβάνουν δεσμεύσει, όλου του είδου τα βήματα συζήτηση, αλλά δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο τι εμπίπτει στου συνολικού στόχου. Α πούμε, στόχο για βελτίωση τη ασφάλεια των τροφίμων, ε, βελτίωση ε, χρηματοδότηση ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματο. Πώς θα βοηθήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια αν δεν είναι και σαφείς οι στόχοι και αν ε, είναι πρόσθετοι ή εντάσσονται οι στόχοι αυτοί στους παγκόσμιου στόχου. Επίση πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις εθνικές αναπτυξιακές ε, στρατηγικές για να υπάρχει συνεκτικότητα και συνέπεια με τη χάραξη των εθνικών πολιτικών. Έχουμε επίσης αύξηση όλων των πηγών ανάπτυξης. Έχουμε βέβαια και εδώ το ζήτημα της ενεκτικότητας. Πολλοί από τους πόρους δεν κατανέμονται ξεκάθαρα στο ίδιο πλαίσιο. Και αυτό οδηγεί σε συζητήσεις για το κατά πόσον μπορεί να είναι αποτελεσματικό το σύνολο της βοήθειας. Θα μπορούσαμε ίσως στη συζήτηση να εμβαθύνουμε σε κάποια από αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο τώρα, Έχουμε μια μακροχρόνια δέσμευση αναλάβει και υπόσχεση στο πλαίσιο ε, των ε, στόχων ε, των οπτυξιακών να έχουμε ένα δίκαιο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και οι εμπορικέ διαπραγματεύσει του γύρου τη Δόχα έπρεπε να εκπληρώσουν το στόχο αυτό. Δεν έχει ολοκληρωθεί όμω ο γύρο τη Δόχα και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά επίμαχα και εκκρεμή ζητήματα. Αν λοιπόν δεν σημειώσουμε πρόοδο και δεν έχουμε καλύτερη αξιοπιστία για την επίτευξη ενός δίκαιου εμπορικού συστήματος, ε, τότε έχουμε, ε, ε, δεν κινδυνεύουμε την όλη πρόοδο. Θα μπορούσε ίσως η προσέγγιση της πρόορης ή πρόμοιμης να βοηθήσει, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει πρόοδος και να δώσει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διαπραγματεύσεις ε, της Ντόχα. Αν όμως, ε, ακόμη και αν δεν θα επιτύχει συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου για όλα τα θέματα. Επίσης, πρόσβαση στην αγορά είναι πολύ σημαντικό, είδος για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Λίγη πρόοδο σημειώθηκε από το 2004 και μετά, σε ό,τι αφορά την αδοσμολόγητη ή χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά. Δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο, τα πράγματα είναι λίγο σταθερά, λίγο ε, αμετακίνητα και το Μάιο στην Κωνσταντινούπολη είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί πρόσβαση στην αγορά και από τι αναψώμενες αλλά από τι αναπτυγμένε και από τις απορρισμένες αναψώμενες χώρες που θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο για να μπορέσει να υπάρξει βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά. Τέλος, πάντα από αυτού, ένα αμφιλεγόμενο θέμα που ίσως σας αφορά και εσάς εδώ, είναι οι γεωργικές επιδοτήσεις που για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη ΣΥΠΑ, χώρες όσα εγγένει. Σχετικά μειώθηκαν μεν, αλλά σε απόλυτους όρους εξακολουθούν να παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Σε ένα επίπεδο τριπλάσιο περίπου. Σε σχέση με το σύνολο της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχεται κάθε χρόνο. Άρα εδώ πέρα αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι πολλές από αυτές τις επιδοτήσεις πλήττουν τα συμφέροντα των αγροτών σε αναπτυσσόμενες χώρες και υπονομεύουν και κάποιους άλλους τομείς που προσπαθούμε να στηρίξουμε με την πολιτική βοήθεια για το εμπόριο ή τις πολιτικές μας για βελτίωση της επιστημικής ασφάλειας. Και αυτό μας δημιουργεί ανησυχία. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα σε όλη την αναπτυξιακή ατζέντα. Για να μην δαπανίσω πολύ από το χρόνο σας θα μιλήσω εν συντομία για την ε, ατζέντα μετά το 2015. Και μετά τη συνεδρίαση ελπίζω να έχετε το χρόνο να εξετάσετε την ίδια την έκθεση. Λοιπόν, ε, για την περίοδο μετά το 2015 έχουμε αρχίσει τις εργασίες στον ΟΗΕ για να οργανώσουμε δηλαδή τις συζητήσεις και στους κόλπους της γραμματείας και με τα ε, κράτη-μέλη. Η έκθεση του Γενικού Γραμματέα στις 18 Νοεμβρίου στη Γενική Συνέλευση θα συζητηθεί και περιέχει ανάλυση της πρόοδου προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετής αλλά καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν για το νέο θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 2015. Ε, χωρίς να προδικάζουμε τις συζητήσεις που θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση, θα σας πω ότι προτείνει αυτή η έκθεση ένα σημείο εκκίνησης, ένα εφαλτήριο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσει το θεματολόγιο να ισχύει για, και μετά το 2015 για δύο λόγους. Πρώτον, ε, το 2015 είναι προθεσμία για να υλοποιηθούν ε, κάποιοι από τους στόχους, αλλά όχι όλοι. Ε, για την φτώχεια θα έχουμε με μείωση κατά 50% σε σχέση με το επίπεδο του 90 ε, μέχρι το 2015 και το ίδιο ισχύει και για κάποιους άλλους ε, στόχους της χιλιετίας. Δεύτερον, φυσικά δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τον πυρήνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, δηλαδή τους ίδιους τους ανθρώπους, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα συνεχίσει να ισχύει αυτό. Ε, πολλοί λένε ότι πριν προχωρήσουμε πρέπει να γίνει συνολικός απολογισμός των, του ωφέλους ε, που προσφέρει ε, το θεματολόγιο με αυτούς τους στόχους της χιλιετίας. Ε, δηλαδή να κάνουμε τη σύγκριση με την κατάσταση όπως θα ήταν αν δεν είχαμε υιοθετήσει αυτούς τους στόχους χιλιετές. Να δούμε δηλαδή τα ωφέλη μιας τόσο ευρεία αναπτυξιακής ατζέντα. Κατόπιν υπάρχουν ζητήματα που εμέσως υπονοούνται δηλαδή στην ατζέντα μετά το 2015 ή και απουσιάζουν. Σας μίλησα προηγουμένως για τις διάφορες διαστάσεις. Δεν υπάρχει ομοιομορφία σε σχέση με την πρόοδο που σημειώνουμε και άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τις ε, ανισότητες, την πρόοδο που σημειώνουν οι διάφορες χώρες. Επίσης ο πληθυσμός, οι νέες ε, τάσεις ε, θα έχουν ιδιαίτερη σημασία, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε επισητιστική ασφάλεια και ασφάλεια των τροφίμων ε, γίνονται ολένα και πιο επιτακτικές ανάγκες να κινηθούμε λόγω της ένδυας ε, των λιμών κτλ. Κλιματικές αλλαγές ε, και κλιματική αηφορία. Αυτό είναι ένα επιμέρους στοιχεία στοιχείο των στόχων της χιλιετίας, αλλά δεν μπορούμε και να υπερβούμε το φυσικό μας περιβάλλον όσο και αν το θέλουμε και στα θα, αυτό θα ε, αποτελεί στοιχείο κλειδί στη νέα ατζέντα. Ε, έλλειψη ειρήνης επίσης ε, είναι ένας βασικός λόγος έλλειψης προόδου προς την επίτευξη των στόχων της χιλιοτίας. Λοιπόν, να δούμε τώρα για τη νέα ατζέντα. Είπαμε ότι θα αρχίσουμε από έναν απολογισμό σε σχέση με την δήλωση της χιλιετίας. Για δείτε λοιπόν τις αρχές που θα διέπουν όλες τις νέες προκλήσεις. Τις... Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε, εκτός και αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να μην το κάνουμε, να επιβεβαιώσουμε τις συμπεφωνημένες αρχές που συναποτελούν την ατζέντα, δηλαδή οι ατομικές ελευθερίες, η συμμετοχική ε, ε, διακυβέρνηση, αυτά συνδέονται με τις προκλήσεις που προανέφερα, ε, ισότητα ανάμεσα στα έθνη και στα άτομα, αλληλεγγύη για να διαχειριστούμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, ανεξιθρησκεία, πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε τους πληθυσμούς και την πίεση από τη μετανάστευση, ε, σεβασμός για τη φύση, για την αηφόρο ανάπτυξη, για ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε σε παγκόσμιο επίπεδο την οικονομική και κοινωνική πρόοδο ε, κάποιοι αναπτυξιακοί στόχοι, βιώσιμοι αναπτυξιακοί στόχοι, μάλλον θα είναι στον πυρήνα της νέας ατζέντα ή ας το πω πιο ήπια, δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε ε, νέο θεματολόγιο που να ε, μην έχει στον πυρήνα της αυτούς τους ε, βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους, ε, γιατί δεν γίνεται πλέον να υπερβαίνουμε τα όρια του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ε, τέλος πάντων και θα ολοκληρώσω τώρα σε λίγο. Οι βασικές προκλήσεις ε, μας έχουν μείνει. Είπαμε ότι η αηφορία θα είναι στον πυρήνα του νέου θεματολογίου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μετά το 2015 χρειαζόμαστε μια πραγματικά αναπτυξιακή ατζέντα. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχο. στόχος ε, με τους στόχους της χιλιετίας και καλό είναι να βοηθούμε τις φτωχές χώρες και τους στόχους, αλλά να επιδιώκουμε βιωσιμότητα στην ανάπτυξη θα πρέπει ε, ε, να ισχύουν αυτά για όλους, για τα ε, πλούσια και για τα φτωχά κράτη, για τους έχοντες και μη έχοντες. Νομίζω ότι σε αυτές τις γραμμές θα πρέπει να υιοθετήσουμε το νέο μας θεματολόγιο. Τι θα χρειαστεί λοιπόν για να επιτύχουμε τους στόχους μας, ποια είναι η διαδικασία. Ε, στη Γενική Συνέλευση θα αναθεωρήσουμε τους στόχους, ε, θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις ε, εντός και εκτός ΟΗΕ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε και τις συζητήσεις μέσα σε αυτά τα πλαίσια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικό το νέο θεματολόγιο φιλόδοξο αλλά ταυτόχρονα εφικτό, υλοποιήσιμο ούτως ώστε οι εκθέσεις που άρχισα να σας παρουσιάζω να είναι όσο το δυνατόν πιο θετικές ε, γίνεται ως προς τα αποτελέσματα. για να έχει μια κοινή ανάπτυξη ολόκληρη οικουμένη. Ευχαριστώ. Τέσσερις ε, συναδέλφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. το όριο τρία λεπτά. Ο κύριος Κάσμαν ε, πρώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μην δώσω τριών λεπτών. Είμαι του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση των στόχων των αναπτυξιακών της χιλιετία. και καλωσορίζω αυτή την έκθεση και την ηγεσία των υπηρεσιών του ΟΗΕ και του Γενικού Γραμματέα του Μπαν Κιμούν ιδιαίτερα. Οι δεσμεύσει στην Σύνοδο και η δέσμευση του Πρόεδρου Μπαρόσο ε, για άλλο ένα δισεκατομμύριο νομίζω πως πρέπει να στηριχθούν και να αναγνωριστούν εάν πρόκειται τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τις υποσχέσεις τους, τις δεσμεύσεις τους για 0,5-0,6% κάτι το οποίο όπως δείχνει το διάγραμμά σας προφανώς δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το Κοινοβούλιο και στην έκθεσή μου και στην έκθεση που θα ψηφιστεί αύριο της ε, κυρίας Ζολή ασχολείται οπωσδήποτε με την συνοχή στην πολιτική που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καθώς η ροή των κεφαλαίων από τις χώρες αυτές ε, υπολογίζεται σε δεκαπλάσια από την αναπτυξιακή βοήθεια καθώς επίσης εκεί όπου εστιάζουμε στην ε, βοήθεια και το πώς θα μπορέσουμε να την ε, διπλασιάσουμε. Αλλά πρέπει βεβαίως να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, αλλιώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. ορίζω επίσης την προσέγγιση για μετά το 2015 και ελπίζω αφού έχουμε θέσει αυτή την ημερομηνία θα δούμε το τι έχουμε επιτύχει. Δεν θα υποχωρήσουμε, ε, δεν θα υποχωρήσει κανένα κράτος μέλος, ε, πολύ περισσότερο οι υπόλοιπε χώρες δωρητές. Οπότε πρέπει να επαναληφθούν οι αρχές του Glenn Eagles και είμαι σίγουρος πως η επανάληψη αυτή βεβαίως ε, μας σημαίνει πως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για αποτελέσματα από τα κράτη-μέλη και τις υπόλοιπες χώρες. Πρέπει να υπάρχει κάποια λογοδοσία. Η Επιτροπή μας νομίζω συμφωνήσαμε πως θα ε, έχει μία ετήσια έκθεση και θα βλέπουμε το τι κάνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τους ε, στόχους τους και πού ε, έχουν μείνει πίσω και όπου έχουν μείνει πίσω θα τις κατονομάζουμε. Και βεβαίως δυστυχώς η αλληλεγγύη δεν είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλες οι κυβερνήσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα. Νομίζω πως μια εικόνα των φτωχών και κατατρεγμένων χωρίς δικαιώματα σε χώρες που δεν είναι μόνο η Αφρική, θα α, μας υπενθύμιζε το τι σημαίνει ελεγγύη. Ελπίζω να τήρησα και τον χρόνο μου, κυρία Πρόεδρε. Απολύτως, ως συνήθως, κύριε Κάσμαν. Κυρία Κέλλερ. Thank you. Um, thank you very much for your Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, η οποία ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και βεβαίω όλοι γνωρίζουμε τις ε, προκλήσεις ε, του 2015 και ίσως να μην λυθούν στο τέλος. Παρ' αυτά, Νομίζω πως καλό είναι να δούμε το τι θα γίνει και μετά το 2015 όπως το κάνατε κι εσείς. Και έχω κάποιες ερωτήσεις. Κάτι το οποίο πάντα ακούμε και από ΜΚΟ όσον αφορά το μετά το 2015 και τι θα κάνουμε είναι μια αδυναμία που θεωρούν ότι υπάρχει είναι πως δεν αναφέρονται το πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι. Μπορεί να τους επιτύχει ο καθένας με όποιον τρόπο θέλει και θα ήθελαν οι ΜΚΟ να δοθεί περισσότερη έμφαση στον τρόπο, παραδείγματος χάρη με μεγαλύτερη συμμετοχή δική τους. Δηλαδή, να μην γίνεται κάτι, παραδείγματος χάρη, ενάντια στέλεση της κοινωνίας των πολιτών και του τοπικού πληθυσμού. Πώς θα λέγατε να συμπεριληφθεί αυτό στην ατζέντα για το 2015 και μετά. Κατόπιν ανησυχώ λίγο για το ότι τώρα μετά το 2015 ή όπως πλησιάζουμε στο 2015 θα πει ο κόσμος ε, δεν πετύχαμε τους στόχους, μπορεί να τους πετύχουμε, μπορεί όχι και μετά οι φιλοδοξίες να μειωθούν ε, σημαντικά για την περίοδο μετά το 2015 για να τεθούν ευκολότεροι στόχοι που θα έχουν μια πιθανότητα να επιτύχουν σε αντίθεση με πολύ φιλοδοξού στόχου οι οποίοι δεν θα επιτευχθούν ίσως. Θεωρείτε πω θα συμβεί. Κάτι τέτοιο θα γίνουν πιο εύκολοι στόχοι ή θα επικρατήσουν αντίστοιχο πνεύμα και θα πούν όχι τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ κύριος Μπέρμαν. Καλό απόγευμα. Ε, έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να μιλήσουμε Ολλανδικά. Ναι, μπορώ. Ωραιότατα. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσίαση αυτή. Καλωσορίζω ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπατε για την ανάγκη του να σκεφτούμε την ανάπτυξη ως ένα δικαίωμα που βασίζεται στα δικαιώματα των πολιτών. Και αυτό ακριβώς βεβαίως ε, γίνεται ε, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι στους στόχους της χιλιετίας. Ελπίζω να ενισχυθεί αυτό στο μέλλον. Αλλά θα ήθελα να σας προσκαλέσω να γίνετε πιο συγκεκριμένος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της. Είστε εδώ πέρα για να μιλήσετε σε εμάς. Θα ήθελα να ε, μας πείτε σε ποιο βαθμό είναι αρνητικές, δηλαδή οι ευρωπαϊκές ε, γεωργικές ε, επιδοτήσεις. Μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Επίσης, να γίνετε πιο συγκεκριμένος πώς η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου είναι αρνητική για τις χώρες αυτές και που πιθανώς όχι, που είναι τα ισχυρά, που είναι τα ασθενή σημεία στην ευρωπαϊκή πολιτική γενικώ. Μιλάμε για συνοχή της πολιτικής για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Θα μπορούσατε να μας τα πείτε αυτά συγκεκριμένα. Δεύτερον, υπάρχει μια φιλία η οποία αυξάνεται στις χώρες αυτές, ε, αλλά και γρήγορη οικονομική ανάπτυξη. Πέντε από τις δέκα πιο αναπτυσσόμενες χώρες είναι στην Αφρική. Θεωρείτε πως η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσαρμοστεί στις γρήγορες αυτές εξελίξεις και τι χρειάζεται γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη, σκέφτομαι εδώ πέρα το πώς θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για να μην αποκλειστεί κάποιος από δάνεια, ασφάλειες, ε, αποταμιεύσεις κτλ. Αυτά θα ήθελα να ακούσω από σας. Ευχαριστώ. Madame Sargentini. Dank u voorzitter. Κύριε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Φώσσα, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας δεν πρέπει να απολογίστε για το ότι μιλάτε πάρα πολύ. Όταν μας λένε επιτέλους εδώ πέρα πως δεν θα επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας, κατά το οποίο δεν είναι ειδήσει, νομίζω πως μπορείτε να μιλήσετε λίγο παραπάνω και να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βέρμαν. Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψτε Σήμερα έχει 10 μήνες, 12 του μηνός η Κομισιόν θα ξεκινήσει το νέο της, ε, την παρουσίαση του νέου της προγράμματος για τη Γεωργία για το 2013 και μετά. Ίσως θα μπορέσετε να είστε παρόν για να παρακολουθήσετε και αυτό επίσης την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τη συνεισφορά του για το ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γύρο της Ντόχας. Έχουμε λοιπόν ένα ψήφισμα το οποίο είναι επικριτικό για ολόκληρο το γύρο και θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα από αυτού και ένα τελευταίο ερώτημα. Το Κοινοβούλιο αυτό κατά την άποψή μου ε, πρόσφατα νομίζω ενέκρινε την πολιτική του Επιτρόπου του κυρίου Ντεχιούχτ για το εμπόριο μέχρι το 2020. Εγώ θεωρώ πως αν υπάρχει μια καλή εμπορική πολιτική δεν χρειάζεται ξεχωριστή αναπτυξιακή πολιτική. Χρειάζεται εμπόριο και αυτό είναι όλο. Οπότε το τι κάνουμε λάθος στην πολιτική μας, την εμπορική και τι μπορούμε να κάνουμε για να προσαρμοστεί η εμπορική πολιτική της Ένωσης για να είναι πιο συνεκτική από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να είστε όπως πάντα σύντομοι σας παρακαλώ. Voilà. Ο κύριος Χαμπέ. Ναι, δεν είχα δει καλά το όνομά σας. Δεν πειράζει, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βος για την παρουσίασή του και για την έκθεση βέβαια, που είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ε, συνεχίζει να ασκεί πιέση σε εμάς ε, ο ΙΕ για να κάνουμε κι εμείς ε, τη δική μας δουλειά σε ό,τι αφορά την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Άκουσα αυτά που είπατε για, τις, για τους στόχους και για το αν τους εκπληρώνουμε ή όχι, αλλά θέλω να σας πω ότι οι δική μας στόχη είναι πολύ πιο φιλόδοξη σχέση με αυτούς που θεσπίζουν άλλοι εταίροι. Σε ό,τι αφορά συνολικά τώρα τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, πιστεύουμε όλοι πια ότι πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να πετύχουμε το 2015 ως το δυνατόν ε, πιο κοντά ε, να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους και ο Μπαρόζο, ο πρόεδρος της Επιτροπής πέρυσι, ξεκίνησε την πρωτοβουλία με ένα δις ευρώ για την ε, στήριξη ε, της προσπάθειας επίτευξης των περισσότερων από τους αναπτυξιακούς στόχους. Ελπίζουμε να αποδώσει καρπούς αυτή η πρωτοβουλία και την επόμενη εβδομάδα η Κομισιόν θα ξεκινήσει την αναθεώρηση της δικής της πολιτικής για την ανάπτυξη ε, υπαίθρου. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Τέλος, σε ό,τι αφορά το θεματολόγιο του 2015, θέλω να σας ευχαριστήσω που μας αναφέρατε τα σχέδια των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπα και εξ αρχής, αυτό που βασικά μας ενδιαφέρει είναι να πετύχουμε το συντομότερο δυνατό του στόχου του 2015. Βέβαια, φυσικά και θα δούμε ε, την περίοδο μετά το 2015 και τι θέματα μπορούμε να λύσουμε από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο για μια ακόμη φορά στον κύριο Βος. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ενθαρρυντικά ε, ερωτήματα που βέβαια ε, αποτελούν και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Σίγουρα ε, δεν νομίζω ότι μπορώ να καλύψω όλα τα ερωτήματα, θα προσπαθήσω τα περισσότερα να τα καλύψω γιατί τα πιο πολλά είναι πολύ σημαντικά, μείζωνα θέματα. Το πρώτο σχόλιο ήταν πόσο σημαντικό είναι να ε, υπάρχει λογοδοσία από όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τους στόχους που έχουν αναλάβει. Έχουμε ανεβάσει και εμείς ε, τον πύχη και ο Γενικός Γραμματέας μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα, τέλος πάντων ένα σύστημα λογοδοσίας μέσω του οποίου πιο συστηματικά θα παρουσιάζουμε τις ελλείψεις, ε, τα κενά, που δεν υπάρχει διαφάνεια, που δεν υπάρχει σαφήνεια σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις. Κάποια από τα αποτελέσματα θα τα έχουμε τον επόμενο μήνα. Θα έχουμε το ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης σε μια πιο σύντομη εκδοχή. και θα είναι μια διαδραστική ιστοσελίδα που θα μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες, να βλέπουν ποιες είναι τι ελλείψεις και αδυναμίες υπάρχουν, τις πληροφορίες που είχαμε και σίγουρα θα είναι ευπρόσδεκτη και η δική σας στήριξη στην προσπάθεια αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημα της κυρίας Κέλλερ τα σχόλια για το ποια θα πρέπει να είναι η φύση του επόμενου θεματολογίου, της επόμενης ατζέντα. Βλέποντας την σημερινή ατζέντα κάποιοι θεωρούν ότι ε, στοχεύει πολύ περισσότερο στους στόχους και όχι τόσο στις διαδικασίες. Αν μπορώ να ερμηνεύσω σωστά το ερώτημά σας κυρία Κέλλερ, συμφωνώ και βέβαια είναι πιο εύκολο διεθνώς να αποφασίσει κανείς ε, μια δέσμη στόχων παρά τον τρόπο επιτευξής τους. Θα πρέπει να δούμε όμως όχι μόνο σαν το στόχους της χιλιετίας. Βλέπετε ότι η ομάδα των 20 των G20 προσπαθεί με τα μεγάλες δυσκολίες να υπάρξει συντονισμός των πολιτικών. Και ακόμη και διμερός ε, είναι αυτό δύσκολο. Άρα πιο εύκολα συμφωνεί κανείς ε, επί των στόχων παρά επί της συγκεκριμένης διαδικασίας και πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί. Συμφωνώ πάντως ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή πρώτα απ' όλα στο βαθμό στον οποίο σημειώνουν οι χώρε πρόοδο προς την επιτεύξη ενό στόχου. Δεύτερον, γνωρίζουμε ότι διαφέρει η κατάσταση από τη μια χώρα στην άλλη. Ίσως αυτό να μην ήταν ο αρχικός στόχος, αλλά τελικά έτσι κατέληξε να βλέπουμε πιο πολύ τους διεθνείς στόχους ε, σαν να είναι εύκολο να εφαρμοστούν οικουμενικά αυτή η στόχη σε όλες τις χώρες. Άρα θα πρέπει να δούμε τα διαφορετικά πλαίσια, να επικεντρωθούμε ε, στα διαφορετικά πλαίσια και στο τι μπορεί να επιτευχθεί και βέβαια τις προσπάθειες για την επιτευχή των στόχων, διότι και από τις δύο άκρες του φάσματος ε, έχουμε προβλήματα. Αν δείτε τις ε, προσπάθειες, αν κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, πρέπει χάρη να μειώσουμε την παιδική θνησιμότητα κατά 50%. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα από 250 να μειωθεί σε 150 ο ρυθμός ε, των ε, παιδιών που πεθαίνουν ή ε, σίγουρα είναι πολύ μεγάλο επίδεμα. Πάτε όμως στις χώρες της Καραϊβικής, αν είναι πολύ μικρή παιδική στις χωρες της Καρυβικής. αν ειναι εκεί και του ζητηθεί να μειωθεί, ακόμα η μεγαλύτερη προσπάθεια θα απαιτηθεί από αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε και σχετικά τι προσπάθειες μπορούν να κάνουν οι χώρες για να σημειώσουν πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Άρα και πάλι πιο εύκολα συμφωνεί κανείς επί των συγκεκριμένων αρχών και όχι επί των τρόπων με τον οποίο κάθε χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ευέλικτοι και αυτό θα φροντίσουμε και για την ατζέντα του 2015. Δεύτερο ερώτημα. Πόσο φιλόδοξα πρέπει να είμαστε. Μήπω πρέπει να φοβόμαστε ότι θα υπάρξει επιβράδυνση των προσπαθειών για την επίτευξη των στόχων του 2015. Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει αυτό ο κίνδυνο, Δηλαδή, αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και αν έχει τρωθεί αξιοπιστία ε, και η φήμη, τότε και η πολιτική και η κοινωνική υποστήριξη μπορεί να χάσει την ορμή που είχε. Άρα, αυτό που πρέπει να γίνει, καταρχά και πάνω απ' όλα, είναι αν συμφωνήσουμε και εξακολουθήσουμε να συμφωνούμε ότι αυτοί οι αξιέπαινοι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν, Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και για μετά το 2015 σίγουρα δικηβεύονται περισσότερα. Αν έχουμε το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, εκεί υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω του φυσικού περιβάλλοντος για το πώς η ανάπτυξη μπορεί να σημειωθεί. Αν μπορούμε να φτάσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, μπορεί να θέσουμε σε κίνδυνο την ανάπτυξη. Άρα οι στόχοι αυτοί πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Αν θέλουμε να έχει μέλλον ο κόσμος μας. Άρα πρώτα απ' όλα χρειάζεται πολιτική βούληση για να συνεχίσουμε και κατά δεύτερον πρέπει να υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε τις προσπάθειες και όλοι έχουμε να κερδίσουμε αν φτάσουμε τα επίπεδα ανάπτυξης που θα θέλαμε να πετύχουμε για όλους. Στους Ολλανδούς συναδέλφους, ε, αλλά θα αναφερθώ ε, σε αυτά που είπαν πάλι μιλώντας αγγλικά, γιατί είναι πιο εύκολο για μένα, για να είναι και πιο εύκολο για τους υπόλοιπους. E Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ε, στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και πού θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον τομέα του εμπορίου, στην ανάπτυξη, γεωργικές επιδοτήσεις, σε ποιο βαθμό είναι επιζήμιες στους αγρότες των αναπτυσσομένων χωρών. Το πιο απλό επιχείρημα κατά των επιδοτήσεων, σίγουρα ε, Μπορεί να δει κανείς το κάθε προϊόν ξεχωριστά, αλλά αν επιδοτηθεί κάποιο προϊόν σε ένα κομμάτι, σε ένα μέρος του κόσμου, δημιουργείται αμέσως ανταγωνισμός. Και υπάρχει ένα είδος ψευδούς, πλαστού ανταγωνισμού τελικά. Οι ε, αγρότες που πρέπει να παραγάγουν αυτό το προϊόν θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα με τον ανταγωνισμό και λόγω των εξαγωγών και λόγω των εισαγωγών, γιατί θα έρχονται τα προϊόντα αυτά, θα εισάγονται στι χώρε του και αυτό θα υπονομεύσει την παραγωγικότητα. Και ίσως αυτό είναι το ισχυρότερο επιχείρημα για την αποφυγή των επιδοτήσεων. Έχουμε το θέμα τη της παραγωγής βάμβακος ε, και ξέρετε στη ΣΥΠΑ τι γίνεται με τους βαμβακοπαραγωγούς στην Κεντρική Ασία, στην Αφρική και γενικά στην Ασία τέλος πάντων. Θα πρέπει όμως τώρα να βρούμε τις σωστές πολιτικές για τη μείωση των επιδοτήσεων και να δούμε πώς μπορούμε να αποζημιώσουμε ίσως τους αγρότες. Δεν μπορεί να γίνει με μια νέα προσέγγιση αυτό και δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εφικτό. Άρα θα πρέπει να στηρίξουμε τους αγρότες μειώνοντας ε, σε τον χρόνο της επιδοτήσεις στις πλούσιες χώρες. Ταυτόχρονα όμως πρέπει η παραγωγική δυνατότητα των αγροτών και άλλων παραγωγών σε αναψώνες χώρες να στηριχθεί. Και έρχομαι σε αυτό που είπε μία από τους ε, βουλευτίνες, ότι δεν είναι μόνο το εμπόριο αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ανάπτυξη, Υπάρχουν μεν ε, κέρδη λόγω του εμπορίου, αλλά αυτά μπορεί να μην είναι και τόσο ορατά σε κάποια μέρη του κόσμου. Το θέμα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη, πιο ισχυρή παραγωγική δυνατότητα στις χώρες, σε διαφοροποίηση της παραγωγικής ικανότητας. Έτσι μπορεί κανείς να αποκομίσει μεγαλύτερο ωφέλη από το διεθνές εμπόριο. Και εκεί η αναπτυξιακή πολιτική μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Το Aid for Trade είναι στο πλαίσιο του θεματολογίου της, ε, ε, του, του ΟΗΕ και το έχουμε ενισχύσει τα τελευταία χρόνια αυτό το δόγμα. Θέλουμε να το ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Το βασικό δεν είναι μόνο για αυτό το πρόγραμμα Aid for Trade να αναθέτονται περισσότεροι πόροι, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές στρατηγικές τι αναπτυξιακές αυτοί ε, οι πόροι, για να βελτιωθεί η παραγωγική δυνατότητα των αντισωμένων χωρών. Τώρα, εμπορικέ διαπραγματεύσεις ε, ίσως ε, να είναι μάταιες, εάν δεν πετύχουμε τους άλλους μας στόχους. Έχουμε κάποιες διμερείς εμπορικές συμφωνίες, περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, χώρες κάνουν πολλέ προσπάθειε για δεσμολόγητη πρόσβαση χωρίς ποσοστώσεις ε, σε αγορές ε, ε, των χωρών που είναι εμπορικοί εταίροι, ακόμη και, πρώτα τα οποία δεν παράγουν. Γιατί λοιπόν, ποιο είναι το νόημα να γίνεται κάτι τέτοιο, όταν δεν, είναι σχεδόν, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου δυνατότητα βελτίωσης της παραγωγικής ικανότητας. Άρα, το ουσιώδες είναι η εμπορική πολιτική και η αναπτυξιακή πολιτική να συμβαδίζουν, να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα σημεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, απαντήσεις της Επιτροπής, με τα χαράς να εξετάσω την αναθεώρηση της αναπτυξιακής, ε, του αναπτυξιακού θεματολογίου, είτε όταν δημοσιευθεί, είτε και νωρίτερα αν μπορέσω να την προμηθευτώ. Και βέβαια για το κατά πόσο θα είμαστε εδώ στο 10 Οκτωβρίου. Όχι, δεν θα είμαστε, θα έχουμε επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. J'invite Grandi à nous rejoindre. Προσέλθετε αν θέλετε στο βήμα κύριε Γκράντι.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 Alors, nous allons continuer notre séance. De... Συνεχίζουμε λοιπόν πάνω από 60 χρόνια δραστηριοποιείται η υπηρεσία του ΟΗΕ ονόματι ο για τους, ε, Παλαιστινια... Ε, για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Ε, βοηθάει εκατομμύρια πρόσφυγες στην Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη, στην Ιορδανία, στο Λίβανο και στη Συρία πέρυσι. Ανήκα σε μια αντιπροσωπεία των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων Προϋπολογισμών και Ανάπτυξης που μετέβει στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη για να συνειδητοποιήσει ποια είναι η κατάσταση επί επιτόπου και να κατανοήσει πώ θα γίνει πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή βοήθεια επιτόπου. Διαπιστώσαμε ότι η Ούνρα ε, ε, επιτελεί εκπληκτικό έργο και ε, πραγματικά συγκινήθηκα από αυτήν την εμπειρία. Ε, στην εποχή της Αραβικής ε, Άνοιξης ε, ζητείται με η θέσπιση η ίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού έτους και εξετάζεται από την 66η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το αίτημα αυτό. Σε αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή καλούμε τον Γενικό Επίτροπο της Ούνερα, τον κύριο Φίλιππο Γκράντι. Καλωσορίσατε. Καλωσορίζω επίσης τους φίλους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με την οποία οργανώνουμε από κοινού τη σημερινή συνάντηση και καλωσορίζω και τα μέλη της Επιτροπής των Προϋπολογισμών που παρίστανται σήμερα. Θα ήθελα να τονίσω επίση ότι την περασμένη εβδομάδα η Επιτροπή των Προπολογισμών επί τη αιτήση των Επιτροπών Ανάπτυξη και Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε μια τροπολογία ω προ τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό του 2012 με στόχο να αυξήσει την γραμμή του προπολογισμού τη UNRWA μέχρι τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Γκράντι, με αδημονία αναμένουμε την παρουσίασή σας για την πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τις γειτονικές χώρες. Ε, κατά τη γνώμη σας, ε, ποιες προοπτικές υπάρχουν για να αλλάξει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με ποιο τρόπο μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ανθρωπιστικές ανάγκες ε, σε αυτή την περιοχή του κόσμου και ποιος είναι ο ρόλος που θα έπρεπε να διαδραματίσει η Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Θα σας δώσω το λόγο για 15 λεπτά. σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ε, σας ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη σημερινή σας ε, συνεδρίαση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, αλλά κάθε φορά μου δίνεται μια σημαντική ευκαιρία να συναντηθώ με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας έχουν υποστηρίξει και συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρουσίαση στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε και μετά θα είμαι στη διάθεση των μελών της Επιτροπής για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Τελευταία φορά που ήρθα στις Βρυξέλλες ήταν ε, πριν από ένα μήνα. Επευκαιρία της υπογραφής μιας κοινή ε, δήλωσης με την ε, Κάθη Άστον και τον Επίτροπο Φίλε μέσω της οποίας ανανεώσαμε την οικονομική μας ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα τρία χρόνια. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο χωρίς καμία αφιβολία έχει καταστήσει δυνατή αυτή την συνεργασία με την οποία βέβαια θεωρούμε πως μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην Μέση Ανατολή χωρίς να είναι πολιτικός αυτός ο ρόλος και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω για τη στήριξή σας αυτή. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σύντομη παρουσίαση των βασικών τομέων εργασίας μας. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο. Ε, εγώ θα έλεγα πως το πλαίσιο στη Μέση Ανατολή έχει καθοριστεί από τρεις κυρίως παράγοντες από την τελευταία φορά στην οποία συναντηθήκαμε. Το ένα είναι αυτό το οποίο λέμε Αραβική Άνοιξη. Δεύτερον, μια στάσιμη διαδικασία ειρηνευτική και τρίτον η απόπειρα των Παλαιστινίων να αναγνωριστούν ως κράτος. Η Αραβική Άνοιξη, η οποία είμαι σίγουρος πως σας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές. Ε, έχει διαφορές πτυχές. Έχει βεβαίως και ευκαιρίες, ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και όπως είδαμε όλοι στην Αίγυπτο τις τελευταίες ημέρες ε, βεβαίως παρουσιάζει και κάποιες προκλήσεις αλλά σε γενικές γραμμές από τη σκοπιά της Μέσης Ανατολής οι άνθρωποι μεταξύ των οποίων ζούμε θεωρούν την διαδικασία αυτή πολύ δυναμική και ως μια ευκαιρία για να διαμορφώσουν το μέλλον. Ρεαλιστικά το βλέπουν, θεωρώ πως ο κόσμος στη Μέση Ανατολή δεν έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες, αλλά σε γενικές γραμμές είναι κάτι που το βλέπουν θετικά. Και σε αυτούς που βλέπουν ε, έτσι την ε, Αραβική Άνοιξη θα ήθελα να συμπεριλάβω και τα 5 εκατομμύρια σχεδόν Παλαιστινίους πρόσφυγες με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Από την άλλη, οι Παλαιστίνοι βλέπουν την Αραβική Άνοιξη σε αντίθεση με την στασιμότητα των πολιτικών διαδικασιών που τους αφορούν άμεσα και ειδικά τη στασιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας και ίσως περισσότερο βεβαίως από όλου οι πρόσφυγες, οι μισοί Παλαιστίνοι δηλαδή που βλέπουν τη διαφορά αυτή ε, της δυναμικής ε, διαδικασίας και της στάσιμης διαδικασίας ε, στην οποία κατά την άποψή τους δεν επενδύει αρκετά η διεθνής κοινότητα για να έχει αποτελέσματα, ειδικά από τη δική τους σκοπιά. Η αντίθεση αυτή είναι ώρες-ώρες δραματική και έχει δημιουργήσει εντάσεις τις οποίες βλέπουμε σε διάφορα μέρη της περιοχής. Όσον αφορά τώρα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, αυτό επίσης μεταξύ των Παλαιστινίων είναι κάτι το οποίο το βλέπουν ρεαλιστικά με όλους τους περιορισμούς που υπάρχουν αλλά και θετικά. Ο πρόεδρος ο Αμπού Μαζέν επέστρεψε στη Ραμάλα ως ήρωας. Η αξιοπιστία του ενισχύθηκε στο εσωτερικό μετά την ομιλία στην Γενική Συνελευθερία θα ήθελα εγώ δεν θα σχολιάσω περισσότερο από αυτό, απλά ορίζει το πλαίσιο, απλά θα ήθελα να κάνω ένα ακόμα σημαντικό σχόλιο προς αυτό. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε, όπως σημειώσαμε και εμείς δημοσίως, πως ανεξαρτήτως του αποτελέσματος αυτής της ε, διαδικασίας, της προσπάθειας αυτής, δεν θα αντιμετωπιστεί έτσι το πρόβλημα των προσφύγων. Το προσφυγικό μπορεί να λυθεί μόνο μέσω μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων που θα αφορά ειδικά τους πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να το πούμε γιατί ακόμα και σε δύσκολα μέρη όπως ε, στο Λίβανο και στην Γάζα ε, βλέπουν θετικά το ζήτημα αυτό οι πρόσφυγες αλλά ανησυχούν για το ότι ίσως γίνει μια ευκαιρία να παραμεριστεί το προσφυγικό ζήτημα χωρίς να ε, έχει την πολιτική προσοχή που αξίζει. Οπότε, από την πλευρά μας, παρά το ότι δεν είμαστε πολιτικός οργανισμός, πρέπει να τονίσουμε πως η Ούνρα, παρά τα όσα έχουν πει κάποιοι, θα συνεχίσει να υπάρχει και να επιχειρεί. Είναι σημαντικό να συνεχίσει να επιχειρεί παντού και στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, μέχρι να επιληθεί το προσφυγικό ζήτημα στο σωστό του πλαίσιο που είναι η ειρηνευτική διαδικασία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για να εστιάσουμε τώρα στις πιο συγκεκριμένες ε, επιχειρήσεις ε, της δουλειάς μας. Βέβαια, η κατάσταση στη Συρία είναι πολύ πολύπλοκη. Έχετε δει τις αναφορές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πολύ ανησυχητικές. Επίσης πρέπει να τονίσω πως ε, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες ε, σε μεγάλο βαθμό έχουν παραμείνει απόντες από αυτή την ε, σύγκρουση που είναι κατά βάση μια ένταση μεταξύ του λαού και της κυβέρνησης. Δεν μπορώ εγώ να πω πως υπάρχει στόχευση των Παλαιστινίων προσφύγων. Υπάρχουν γύρω στις 500.000 στη Συρία, αλλά αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι πως οι Παλαιστινοί πρόσφυγες όπως και ο υπόλοιπο πληθυσμός Βεβαίω, κατά καιρού βρέθηκαν μεταξύ των πυρών και έχουν ε, υποφέρει από την καταστολή των διαδηλώσεων. Υπήρχαν περιπτώσεις στην Ντέρα, στον Νότο, στην χόμ στο κέντρο της χώρας. Η πιο κραυγαλαία περίπτωση ήταν στη Λατάκια, στις ακτές όπου η καταστολή της κυβέρνησης συμπεριέλαβε βεβαίω και ένα προσφυγικό στρατόπεδο. Οι πιο πολλοί εκτοπίστηκαν, αλλά τώρα έχουν επιστρέψει και κάποιοι δυστυχώς σκοτώθηκαν. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως δυστυχώς εάν συνεχιστεί η σύγκρουση έχουμε περισσότερα επεισόδια με Παλαιστινίους ε, πρόσφυγες. Ε, γιατί βεβαίως οι περισσότεροι από αυτούς ζουν ε, μέσα και γύρω σε πόλεις και μέσα και γύρω από τις πόλεις γίνονται οι διαμαρτυρίες. Δυστυχώς λοιπόν μπορεί να επαναληφθούν αυτά τα γεγονότα. Η Ούνρα θα παρακολουθεί την κατάσταση. Δεν έχουμε εντολή να σχολιάζουμε βεβαίω την κατάσταση, αλλά οπωσδήποτε θα συνεχίζουμε να υψώνουμε τη φωνή μας όταν επηρεάζονται Παλαιστινοί πρόσφυγες από την εσωτερική αυτή κατάσταση. Και θα κάνουμε δημόσιες δηλώσεις εάν αυτό χρειαστεί. Η ανθρωπιστική αποστολή του ΟΗΕ που επισκέφθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στη Συρία, όπως γνωρίζετε, δήλωσε πως δεν υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Το ζήτημα είναι ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι μια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεγάλων διαστάσεων. Συμφωνούμε με αυτό, παρά το ότι υπήρχαν κάποιες εστίες ανθρωπιστικών προβλημάτων που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Υπήρχε κάποιοι χάναν τη δουλειά τους γιατί... λόγω της κατάστασης. Προσπαθήσαμε με διανομή μετρητών στους πιο ευάλωτους να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Επευθύναμε μια έκκληση για 8 εκατομμύρια δολάρια και είχαμε κάποιες ήδη δωρεές. Στο Λίβανο βεβαίως η ανησυχία είναι πάντα πως οι ταραχές στη Συρία μπορούν να εξαπλωθούν και εκεί πέρα και να προσταθεροποιήσουν μια χώρα η οποία έχει παραμείνει περιέργως σταθερή στους τελευταίους μήνες, αλλά ε, ξέρετε πως ε, κατά βάση είναι μια εύθραυστη χώρα και μέλος βεβαίως της, ε, του εύθραυστου αυτού χαρακτήρα οφείλεται στα 12 περίπου στρατόπεδα Παλαιστινίων προσφύγων όπου οι συνθήκες είναι άθλιες και άρα εκεί πέρα υπάρχει κίνδυνος ταραχών προβλημάτων όσον αφορά την ασφάλεια, εξτρεμισμού και γενικώ εκμετάλλευσης της στόχιας. Γι' αυτό είναι σημαντικό, πρέπει το πούμε αυτό, το ότι λάβαμε πρόσφατα μέσω του μέσου σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαντική χρηματοδότηση για να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες διαβίωσης στο Λίβανο. Αυτή η συνεισφορά δεν είναι μόνο σημαντική για αυτούς που θα υποφετληθούν από αυτήν όσον αφορά τις υποδομές, στέγαση κτλ. αλλά και ως μια σημαντική, αν και μικρή συνεισφορά για σταθεροποίηση μιας ε, ευάλωτης πλευράς ε, της Ιορδανίας. Του Λιβάνου, με Η Ιορδανία είναι ίσως η πιο σταθερή από αυτές τις χώρες, αλλά και η Ορδανία έχει κάποια ευαίσθητα ευπαθή σημεία τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως είναι σε επαγρύπνηση. Η Ορδανία ανισχύει για την στασιμότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας και δικαίω θεωρούν πως ε, έχουν κάποιο ενδιαφέρον στα ζητήματα του τελικού καθόλου, χρήση του νερού, η ε, Ιερουσαλήμ και βεβαίω οι πρόσφυγες, 2 εκατομμύρια πρόσφυγες ζουν στην Ιορδανία, σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας. Η UNRWA επιχειρεί στην Ιορδανία, είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το κράτος. Μιλάμε για 7.000 Παλαιστινίους στους οποίους απασχολούμε και άρα μπορώ να σας ενημερώσω με ικανοποίηση πως η κυρία Άστον προσεκάλεσε την UNRWA να αποτελέσει μέρος της δύναμης εκείνης της ομάδας δράσης η οποία θα συνεχίσει και θα ξεκινήσει εργασία σε λίγες εβδομάδες και χαιρόμαστε για την αναγνώριση αυτή, για το ότι θα μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της Ιορδανίας και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας στηρίξει στο ρόλο μας αυτό. Για να έρθω τώρα στο βασικό θέμα που μας απασχολεί βεβαίως ε, τα, τις καταχώμενες περιοχές. Όπως είπα, ο πρόεδρος Αμπάς ήρθε στην Ραμάλα έχοντας κερδίσει στήριξη από τον λαό του, αλλά βεβαίως διακυβεύονται πολλά για αυτόν αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό το οποίο θα συμβεί στη συνέχεια, εάν θεωρηθεί αποτυχία, μπορεί να οδηγήσει σε ταραχές. Αν ε, βεβαίως εξαρτάται και από το πώς θα εξελιχθεί αυτό. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ταραχές. Ξέρετε, είχαμε πρόσφατα τις δηλώσεις, την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ε, να επεκτείνουν ε, και άλλο τις, ε, τους επικισμούς με την έγκριση άλλων 1.100 κατοικιών και κάποιες πληροφορίες οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν για το ότι κάποιοι στους οικισμούς είναι οπλισμένοι και έτοιμοι να αντισταθούν. Η αύξηση των κατεδαφίσεων των σπιτιών, είδαμε μεγάλη αύξηση στις κατεδαφίσεις, έχουμε τα νούμερα αν θέλετε, ε, πλέον να σας δώσω μια αίσθηση, 42% αύξηση των κατεδαφίσεων σε σύγκριση με το 2010 από την αρχή αυτού του έτους. Όλα αυτά τα στοιχεία ε, προκαλούν βεβαίως ένταση. Ειλικρινά ανησυχώ πάρα πολύ για το ότι εάν υπάρξει ένα επεισόδιο π.χ. κοντά σε έναν οικισμό, είναι τόσο τεταμένη η κατάσταση που μπορεί να κλιμακωθεί πάρα πολύ γρήγορα και είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε σε Παλαιστινίους και Ισραηλινούς την ευθύνη τους για να διατηρήσουν την κατάσταση όσο δυνατόν πιο σταθερή. Από την άλλη στη Γάζα, και θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ πέρα ακόμη μια φορά, το εξή ο αποκλεισμό της Ισραηλινής κυβέρνησης από το 2007 έχει χαλαρώσει, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε αυτό. Μπορέσαμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή κάποιων έργων ανοικοδόμησης, αλλά αποκλεισμό εξακολουθεί να υφίσταται και νομίζω πως είναι σημαντικό και ξέρω πως το έχει κάνει το Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε στους πάντες πως ο αποκλεισμό αυτός αντιβαίνει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και στα δικαιώματα του λαού της Γάζας και άρα θα πρέπει να αρθεί τούτου λεκθέντος βεβαίως εκτιμούμε πως ε, πρόκειται για μια διαδικασία πολύπλοκη και εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει κάνει η Ισραηλινή κυβέρνηση για να διευκολυνθεί η διέλευση κάποιων αγαθών που είναι απαραίτητα ειδικά οικοδομικά υλικά για τα πολλά έργα ανοικοδόμησης που πρέπει να γίνουν. Η οικονομία συνεχίζει να είναι το βασικό πρόβλημα η ανεργία υπάρχει αλλά έχει μειωθεί λίγο γιατί βεβαίως η ανοικοδόμηση δημιουργεί δουλειέ. Η ανεργία λοιπόν εκτιμάται πως είναι στο 33% ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο και η δυναμία εξαγωγής από τη Γάζα στο Ισραήλ και στη Δυτική Όχθη που παραδοσιακά ήταν οι βασικές τους άγορες σημαίνει πως ο ιδιωτικός ε, τομέας ε, μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέσω των τούνελ, δηλαδή παρανόμως ή σε γενικές γραμμές ο πληθυσμός μπορεί να ε, ωφεληθεί από μισθούς που πληρώνει η Ούνρα ή η Παλαιστινιακή Αρχή κατά βάση με ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε η οικονομία που υπάρχει στη Γάζα είναι τεχνητή, είτε είναι επιδοτημένη είτε παράνομη. Η κανονική οικονομία που θα βασίζεται σε έναν υγιή ιδιωτικό τομέα και αυτό είναι δυνατόν να γίνει στην Γάζα γιατί είναι πολύ επιχειρηματικοί άνθρωποι, έχει τελείως καταπνιγεί μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού. Ο μηχανισμός επίσης έγκρισης των έργων ε, και έχει βελτιωθεί και συζητάμε με τον Ισραηλινό στρατό πρέπει να επιταχυνθεί αλλιώς χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να γίνει κάποια ανοικοδόμηση. Όσον αφορά τώρα την ούνρα συνολικά, πάντα μου λένε πως ε, τον ε, διατηρείται η ούνρα σε λειτουργία δεδομένης της ε, ειρηνευτική διαδικασία φαίνεται πως θα χρειαστεί να λειτουργεί η ούνρα είναι κάτι το οποίο κοστίζει πάρα πολύ για τη διεθνή κοινότητα. αυτό είναι αλήθεια. Αν προσθέσει κανείς όλη τη χρηματοδότηση που έχουμε φτάνουμε πάρα πολύ γρήγορα στο 1 εκατομμύριο, δισεκατομμύριο ευρώ το έτος. Αυτό είναι το κόστος ε, λειτουργίας της Ούνρα. Αλλά εγώ πάντα λέω πως αυτό δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο ως κόστος μιας επιχείρησης, αυτό είναι το κόστος μιας πολιτικής αποτυχίας. Έτσι πρέπει να το δούμε. Μόνο εάν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στη ρίζα του, στη, στο πολιτικό επίπεδο μπορεί να ελαφρύνει αυτό το κόστος για τους φορολογούμενους στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και αλλού. Και γι' αυτό και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο όταν έχει τελματωθεί η ειρηνευτική διαδικασία. Βεβαίω, εμείς προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί οικονομικά. Είμαστε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου και προσπαθούμε να μοιραστούμε το βάρος. Είχαμε κάποιες επιτυχίες με Άραβες δωρητές. Η Σαουδική Αραβία φέτος ε, ήταν η τρίτη μεγαλύτερη δωρητή στον ΟΝΡΑ, σύνολο του περιπολογισμού, οπότε σημειώνεται κάποια πρόοδος, αλλά εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ε, αν δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι, ο κόσμος υποφέρει και η ούνρα επίσης εκτίθεται και στους κριτικούς της. Υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν επιτόπου στη Γάζα, στο Λίβανο ιδιαίτερα που έχουν συμφέρον στο να αποδυναμώσουν την Ούνρα. Ξέρετε πως είχαμε διάφορες ευκαιρίες ε, χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή η πιο δραματική έλλειψη κονδυλίων είναι Περιέργως στην Γάζα, όπου δεν είχαμε στο παρελθόν προβλήματα. Τα προγράμματα ε, που αφορούν ψητιστική βοήθεια, δημιουργία, θέσεων εργασίας και άλλες ανθρωπιστικές δραστηριότητες ε, δεν έχει κονδύλια, αλλά και ο βασικός μας προπολογισμό βεβαίως ε, είναι πάντα δύσκολος. Δηλαδή δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε μισθούς δασκάλων, γιατρών, όλων των υπηρεσιών που παρέχουμε κατά και οι μισθοί τους οποίους πληρώνουμε εμείς ε, υπολογίζονται με βάση τους ε, μισθούς του δημοσίου στις χώρες στις οποίες φιλοξενούμαστε. Και ξέρετε πως οι χώρες στις οποίες φιλοξενούμαστε ε, αυξάνουν τους μισθούς του δημοσίου υπό την πίεση της Αραβικής Άνοιξης. Οπότε πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε. Και αυτό για εμάς είναι απαγορευτικό κόστος. Αλλά εάν δεν ε, δώσουμε αυτές τις αξίες τότε υπάρχουν ταραχές. Ακόμα και απεργίες. Ε, από τους δικούς μας έχουμε 13.000 υπαλλήλου στη Μέση Ανατολή. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλος εργοδότης, οπότε η έκκλησή μας είναι να αντιληφθούν τη συγκεκριμένη κατάσταση οι δωρητές και να στηρίξουν την βασική μας χρηματοδότηση, αλλά όπως είπα, όπως είπε η Πρόεδρος, χαιρόμαστε για το ότι υπάρχει θετική απάντηση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ξέρετε, η κοινή δήλωση που υπέγραψα με την Κάθη Άστον και τον Στέφα Φιούλε πριν από ένα μήνα αύξησε τη βασική μας χρηματοδότηση από τα 66 στα 80 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ούνρα το έτος. Και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε μια έκτακτη περαιτέρω συνεισφορά για φέτος που ελπίζω πως θα γίνει πριν το τέλος του έτους. Είναι σημαντικό αυτό για να βγει ο χρόνος. Πρόκειται για τη βασική μας χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε και τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να διατηρήσει την βοήθεια στους Παλαιστινίους γενικώ, όχι μόνο στην ΟΝΡΑ, σε υψηλό επίπεδο. Εμείς θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδώσει και αυτό ειδικά σε καιρούς ε, αβεβαιότητας με τις ΗΠΑ όχι τόσο πολύ για την Ούνρα, αλλά με την Παλαιστινιακή Αρχή. Επίσης θα θέλαμε να σας πενθυμίσουμε πως έχει κρίσιμη σημασία πως το μερίδιο της Ούνρα να συνεχίσει να είναι ανάλογο και επαρκές και βέβαια κρίσιμη σημασία έχει και θέλω να σας το υπενθυμίσω και αυτό πως ε, οι Παλαιστίνοι οι πρόσφυγες και όχι μόνο οι Παλαιστίνοι γενικώ να αποτελούν τμήμα της στρατηγικής σας, των δηλώσεών σας, των ψηφίσματων σας όσον αφορά την πολιτική της νότιας γειτονίας στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα ξεκινήσει το 2014 ειδικά σε μια στιγμή κατά την οποία ναι περισσότεροι πόροι πηγαίνουν στην Νότια Μεσόγειο αλλά όπου και υπάρχει ανταγωνισμός για αυτούς τους πόρους. Ε, θα απαιτηθούν από την Λιβύη, Αίγυπτο, την Ισία και αλλού. Οπότε γι' αυτό χαίρομαι για το ότι θα είμαστε στην ομάδα δράσης ε, την Ιορδανική γιατί νομίζω πως έχουμε κάποιο ρόλο να παίξουμε εκεί πέρα. Να ολοκληρώσω υπενθυμίζοντάς σας πως 5 εκατομμύρια σχεδόν ε, πρόσφυγες ε, είναι ένα σημαντικός πληθυσμός στη Μέση Ανατολή. Αισθάνονται απομονωμένοι μετά από τρεις γενιές άλυτων προβλημάτων. Η Ούνρα είναι ένα από τα λίγα σημάδια για το ότι η διεθνή κοινότητα δεν έχει ξεχάσει αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό είναι σημαντικό να συνεχίζετε να μας στηρίζετε. Οργανώνουμε το Μάρτιο του 2012, 19 και 20 του μηνός, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια εκδήλωση εδώ στις Βρυξέλλες, για να παρουσιάσουμε το έργο μας και να παρουσιάσουμε επίσης τη συνεργασία μας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά θα είναι ε, ε, μια εκδήλωση υψηλού επίπεδου που θα είναι και σε άλλους διεθνείς φορείς. Είναι σημαντικό λοιπόν και ελπίζουμε να παρευρεθούν σε δυνατόν περισσότεροι ευρωβουλευτές για να στηρίξουν την εκδήλωση αυτή. Και εδώ πέρα, κυρία Πρόεδρε, ε, θα ολοκληρώσω. Σας ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τους βουλευτές τώρα. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί υπερβήκαμε κατά πολύ το χρόνο μας. Ε, κύριε Ντέβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γκράντι. Πολύ καλή ήταν η παρουσίαση της κατάστασης. Έμαθα πως ένα από τα ζητήματα στην περιοχή αυτή είναι το νερό. Ε, το πόσιμο νερό, ε, ο καθαρισμός των λιμάτων. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε ε, περισσότερο πόσιμο νερό, κυρίως στα παιδιά, στα πλαίσια της βοήθειάς μας. Θα μπορούσαμε επίσης ε, να βοηθήσουμε ε, αυτά τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα ψυχοκοινωνικά τραύματα που έχουν βιώσει λόγω της βίας που επικράτει στην περιοχή. Έχω και άλλη μία ερώτηση. Νομίζω θα μπορούσε να μας το διευκρινίσει ο κύριος Γκράντι. Άκουσα καλά, είπατε ότι είναι ένοπλοι πλέον οι έπικοι και ότι έχουν τη δυνατότητα να σκοτώνουν στην περιοχή αυτή. Άκουσα καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριος Βέγγελ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Γκράντι, πάντοτε με χαρά ε, παρακολουθούμε την παρουσίαση των εκθέσεων του οργανισμού σας. Ε, είμαστε ευγνώμονες, διότι ήσασταν σαφέστατος και ταπεινόφρονος στην παρουσίαση που μας κάνατε. Σε αυτή την περιοχή του κόσμου όπου είναι πραγματικά κέρια σημασία ο ρόλος της ούνερας. Χαρητήρια για το έργο σας. Σίγουρα ε, η Ούνρα είναι βασικός ε, πολιτικός παίκτη ε, στην Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται για μία ακόμη ανθρωπιστική οργάνωση. Είτε θέλει κανείς να το παραδεχτεί, είτε όχι. Ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή την παράθεση όλων αυτών των γεγονότων που μας αποκαλύπτεται καθώς και την εκτίμησή σας και την άποψή σας για την κατάσταση. Μα μιλάτε για τις προσπάθειες που κάνει η όνορα στη Γάζα επίσης. Είναι συναρπαστικό πιστεύω το πώς υπό αδύνατες ουσιαστικά συνθήκε. τονώνεται την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων εκεί και η αυτή απόδειξη είναι τα, οι θερινοί αγώνες για τα παιδιά είναι φανταστικό, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για το έργο σας. Ε, μπορώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Μπορεί να θεωρήσετε ότι είμαι προκλητικός, αλλά αυτό πιστεύω. Θα ήταν τόσο καλό αν έπαιζαν και παιδιά από το Ισραήλ σε αυτούς τους θερινούς αγώνες ε, της ε, Λωρίδας της Γάζα θα ήταν ευίωνο για το μέλλον, θα αναπτέρωνε το, τις ελπίδες μας. Επίσης ε, θέλω να συμμεριστώ το φόβο σας ότι μας είπατε ότι φοβάστε ότι θα παραταθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η παρουσία σας εκεί παρότι το απέφιαστε. Η πολιτική κατάσταση δεν είναι πολλά υποσχόμενη. 47 10% αύξηση των κατεδαφίσεων αναφέρατε. Δηλαδή κατά 27% υπερβολικά υψηλό το ποσοστό είναι σκανδαλώδες, ε, είναι ε, ε, πελώριος αυτός ο αριθμός, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Το ίδιο και για το τον αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζα είναι παράνομο, είναι απάνθρωπο, παραβαίνει το διεθνές δίκαιο, είναι παράλογο. Ε, και όλοι θα πρέπει να είμαστε απειδισμένοι με αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει εκεί και με αυτά που διαβάζουμε στην έκθεσή σας Ε, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν πρέπει κανείς να θεωρεί ότι είναι φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν ε, στη Λωρίδα της Γάζας. Με κοιτάζει πολύ επικριτικά η αγαπητή μας ε, ε, προεδρεύουσα. Θα ήθελα να διακόψω εδώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βάγγελ. Ο κύριος Ντερός έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκράντι που ήρθε να μας μιλήσει. Νομίζω ότι η σχέση μεταξύ Ούνρα και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά σημαντική. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερο την Ούνρα και το έργο το οποίο επιτελεί θεωρώ ότι είναι μια από τι μεγαλύτερε επιτυχίε του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε που παρέχει στου πρόσφυγε σε όλη την περιοχή. Γιατί υπάρχουν πολλέ γειτονικέ ε, χώρε και πραγματικά το έργο που επιτελεί εκεί η Ούνδρα είναι εξαιρετικό. Και πρέπει σίγουρα να τις παράσχουμε ώστε να τον μεγαλύτερη υποστήριξη. Το θέμα της διατήρησης της αξιοπιστία της Ούνρα πράγματι είναι άκρο σημαντικό για την περιοχή αυτή. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν στην Ούνρα τους απαιτούμενους πόρους για να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της. Είμαστε ε, την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα ε, στην προσωπία της σχέσης με την ε, Παλαιστίνη είχαμε μια περιγραφή πάρα πολύ ζωφερή για τους επόμενους μήνες σε ό,τι αφορά την ανεπάρκεια των πόρων. 36 εκατομμύρια λείπουν ...220.000 παιδιά δεν δεν έχουν εξασφαλίσει τρόφιμα στην, ε, ε, στα σχολεία και πάρα πολλά δεν έχουν λάβει την, ε, το μερίδιο τροφής για το επόμενο τρίμηνο. Μιλάτε για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ούνερα. Για αύξηση της χρηματοδότησης από 66 σε 80 εκατομμύρια. 100 λέει ο μιλητής. Αυτό θα ε, βρεθεί κάποιος τρόπος να καλυφθούν αυτά τα 36 εκατομμύρια τα οποία ε, υπολείπονται. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέζ, θα είναι τελευταία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω, σήμερα γίνεται μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών εδώ στις Βρυξέλλες. Και στην για διάταξη βρίσκεται το Παλαιστινιακό. Αν κατάλαβα καλά δεν υπάρχει συνένεση μεταξύ όλων των Ευρωπαίων Υπουργών. Και μου θύμισε η συνάδελφος ιδίω τον ρόλο του Ολλανδού Υπουργού στο θέμα αυτό. Τι περιμένετε σήμερα από το Συμβούλιο Υπουργών, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω καλά το όνομα. Κόμψ, κυρία Κάμψ, σωστά το προφέρω. Και εμείς με πολύ μεγάλη χαρά ακούμε πάντοτε τον κύριο Γκράντι να παρουσιάζει και να επεξηγεί τα προβλήματα γιατί και εμείς στην Κομισιόν έχουμε ε, θέμα με τον προπολογισμό και πώς πρέπει να τον κατανείμουμε μεταξύ των διαφόρων ε, ενδιαφερομένων φορέων διότι δεν είναι μόνο η UNRAP έχουμε και την Παλαιστινιακή Αρχή. Και επίσης πάντοτε είμαστε γνώμονες που το Κοινοβούλιο πιέζει να μας βοηθήσει, να έχουμε λίγο ε, μια καλύτερη πρόπτικη για τον προϋπολογισμό και τι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα με τους διαθέσιμους πόρους. Πάντοτε προσπαθούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Δυστυχώς όμως έχουμε μόνο τα χρήματα που έχουμε στη θέση μας και Άρα και για μας αυτό συνιστά μια δυσκολία. Πάντως κύριε Γκράντι θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά γιατί δώσατε πάρα πολύ σαφείς ε, εξηγήσεις και περιγράψετε πολύ ξεκάθαρα την κατάσταση επιτόπου. Ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, έχω και την ε, κυρία Σάμπεβα. Δεν ξέρω, θέλετε το λόγο? Όχι. Όχι. Θα ξαναδώσω τότε το λόγο στον ε, κύριο Γκράντι για να απαντήσει στα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω πολύ γρήγορα. Ίσως το πιο πολύπλοκο ερώτημα ήταν αυτό της κυρίας Γκρέζ. Όπως είπα, η Ούνρα πράγματι είναι ένας παίκτη. Ο ρόλος μας είναι ανθρωπιστικός, παρέχουμε υπηρεσίες Άρα δεν εμπλεκόμεθα στην πολιτική συζήτηση, αλλά τώρα τι περιμένω εγώ από τους πολιτικούς ε, φορείς. Αυτό που περιμένουμε είναι μια αποφασιστική δράση εκ μέρους τους για να επιληθεί η κρίση και να έχει ένα αίσιο πέρας. <coughs> και βέβαια περιμένουμε να τεθεί ξανά επιτάπητο στο θέμα των προσφύγων και να τεθεί επιτάπτως κατά τρόπο που να αναγνωρίζεται να αναγνωρίζονται και οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες των προσφύγων και όχι μόνο να γνωρίζονται το πολιτικό συμφέρον, τα πολιτικά συμφέροντα των πολιτικών πρωταγωνιστών. σω να ακούγεται τοπικό, αλλά μετά την ε, έναρξη της Αραβικής Άνοιξης ίσως να ακούγεται λιγότερο ουτοπικό. Τίποτα πια ε, δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς πλέον ε, τις επιθυμίες των λαών, ούτε τις επιθυμίες των Παλαιστινίων, ούτε τις επιθυμίες των Παλαιστινίων προσφύγων. Βέβαια δεν μπορώ να προκαταλάβω ούτε να προδικάσω τι θα συμβεί στο Συμβούλιο Υπουργών, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κινηθούν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να παίξει ένα πιο αποφασιστικό πολιτικό ρόλο αφού υπάρχει στασιμότητα, υπάρχει τελμάτωση. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να ε, καλύψει τον κενό αυτό χώρο που πιστεύω έπρεπε να είχε καλύψει πολύ νωρίτερα, με επιτρέπετε, αλλά πρέπει πλέον να καταλάβει αυτή τη θέση. Θα πρέπει όχι μόνο να υπάρξει ειρήνευση μεταξύ των διαφορών μερών, αλλά χωρίς ενθάρρυνση, χωρίς πίεση δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνευση. Και αν δεν υπάρχει ειρήνη δεν λύνονται τα προβλήματα που σας περιέγραψα. Πρέπει να συνεχίσουμε όχι απλά να υπάρχουν, αλλά να είμαστε και πιο σοβαροί για το λαό επιτόπου και βέβαια με τον τρόπο αυτό γινόμαστε και ένα επιπλέον βάρος οικονομικό για εσάς όσο περισσότερο είμαστε εκεί στην περιοχή. Τώρα, πράγματι το νερό κύριε Ντέβα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς δεν ε, συμμετέχουμε τόσο πολύ σε προγράμματα σχετικά με τα ύδατα. Απλά κυρίως ε, ε, σε ό,τι αφορά τους καταβλισμούς, το 1 τρίτο των προσφύγων, οι πιστοχότεροι κύριοι, συνήθως ζουν σε καταβλισμούς. Εμείς κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και στη Γάζα και στο Λίβανο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ε, παροχή πόσιμου νερού. Καλό θα ήταν να βρεθούν πόροι για την βελτίωση της ποιότητας του νερού. Στη Γάζα αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη υποβάθμιση των υποδομών και έχει να κάνει με τον αποκλεισμό κατά κύριο λόγο. Στο Λίβανο οφείλεται στο ότι είναι τόσο περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένη η μια από τις ίδιες τις πολιτικές στο Λίβανο που αποκλείουν ουσιαστικά τους μετανάστες, τους πρόσφυγες μάλλον ε, και γι' αυτό είμαστε σε διάφορα επίπεδα για να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι πρόσφυγες και να πάψει ο αποκλεισμό τους ώστε η βελτίωση των υποδομών να ωφελήσει όχι μόνο το γενικό πληθυσμό αλλά και τους πρόσφυγες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Πράγματι, ιδίω σε, μέρη όπω η Γάζα, όπου τα παιδιά έχουν υποφέρει τα μάλλα, όχι μόνο από την απομόνωση λόγω του αποκλεισμού, αλλά και από τι επανειλημμένε στρατιωτικέ εισβολέ ε, που έχουμε συνεχώ λόγω του γενικότερου πλαισίου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή την ψυχοκοινωνική υποστήριξη που ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Όπως είπε όμως και ο κύριος Δερόσα δυστυχώς οι παρεμβάσεις αυτές είναι μεταξύ των παρεμβάσεων που δεν έχουν την επαρκή χρηματοδότηση. Αυτά τα 36 λοιπόν εκατομμύρια που θέλουμε, αν αυτά τα επιπλέον δεν τα βρούμε, Ίσως χρειαστεί δυστυχώς να αναστείλουμε το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής ε, υποστήριξης που είναι πολύ ευεργετικό για τα παιδιά της Γάζας και είναι κρίμα αυτό αν ληφθούν υπόψη και επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα τελευταίο για, τις, ε, ε, για τους σπόρους για τη Γάζα. Όχι κύριε Ντερός, αυτό το οποίο δυστυχώς, έχουμε, μάλλον αυτό το οποίο έχουμε διαπραγματευτεί τα τελευταία χρόνια είναι να έχουμε όθηση των κύριων δραστηριοτήτων στον κύριο προπολογισμό, δηλαδή σχολεία, υγεία, ε, ανακούφιση της φτώχειας. Αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε για τη Γάζα είναι τα έκτακτα ανθρωπιστικά προγράμματα. Έκτακτο ανθρωπιστικό πρόγραμμα που διαρκεί όσο διαρκεί ο αποκλεισμό. Γιατί το προκαλεί η κατάσταση. Μιλάμε για τη διανομή τροφίμων, ε, διατροφή στο σχολείο, ψυχική υγεία, δημιουργία θέσεων απασχόληση δεν θα έχει επιπλέον πόρους ε, μέσω της κοινή δήλωσης αυτό το πρόγραμμα. Συνήθως το πρόγραμμα αυτό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργανά ε, χρηματοδοτείται από το γραφείο ΕΚΟ, αλλά και ο προπολογισμό του ΕΚΟ, όπως ε, είπε και η πρόσωπα της Κομισιόν, λόγω έλλειψης, πόρων από την πλευρά της Κομισιόν και εκεί έχουμε περικοπές. Η Επιτρόπος Γεωργίευα στηρίζει, στηρίζει πάρα πολύ το έργο μας, αλλά προσπαθεί και αυτή να τραβήξει όσο μπορεί ε, αλλά οι πόροι είναι περιορισμένοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάντως όλους ε, για τις ε, εκφράσεις υποστήριξη προς το έργο μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Γκράντι. Ευχαριστούμε θερμά για το πολύ σαφές, σημαντικό μήνυμα που μας δώσατε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα στηρίξει, όπως ήδη στηρίζει, το πολύ σημαντικό έργο της οργάνωσής σας και βέβαια ελπίζουμε να σας δούμε και πάρα πολύ σύντομα ξανά στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε αυτό που είπε ο κύριος Βάγκελ ότι τα παιδιά ε, από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μια μέρα θα μπορούν να παίζουν μαζί. Ελπίζουμε αυτό να είναι πραγματικότητα στο μέλλον. Ευχαριστώ. la réunion est terminée. Εδώ λοιπόν λίγη η συνεδρίασή μας και θα συνεδριάσουν αύριο συντονιστές το πρωί στις 9 και η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ θα συνεδριάσει στις 10 στην αίθουσα αυτή, έτσι δεν είναι, ναι, ωραία. Καλό σας βράδυ. Merci faut pas À bientôt, hein, peut-être euh, peut-être